Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το und der Kommission zu den Schlussfolgerungen der Tagung. είναι η δήλωση για την συνέδριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το λόγο θα πρέπει να πάρει ο κύριος Φαν Ρομπόη, αλλά απουσιάζει. Άρα πρέπει να τον περιμένουμε.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 και εγώ μπορώ να σας διηγηθώ διάφορα για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, άμα θέλετε να ακούσετε δικά μου σχόλια, αλλά... Α, ωραία, ωραία, ωραία. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Είχαμε ξεκινήσει τη συνεδρίαση και έχετε το λόγο Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1η και 2η Μαρτίου ήταν θετική και δεν ε, καλύπτεται από μια άμεση κρίση. Δεν μπορούμε βέβαια να αισθανθούμε ικανοποιημένοι με την αντιμετώπιση των τεράστιων οικονομικών ε, προκλήσεων που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Συνεχείς προσπάθειες σε πολλά ε, μέτωπα παραμένουν απαραίτητες. Το ένα μέτωπο είναι η οικονομική εμπαχίωση, το άλλο είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Πολλοί λένε ότι τα δύο αυτά είναι αντιφατικά. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να μην είναι. Από τη δεκαετία του 30 η κύρια αντίδραση στην ε, οικονομική ύφαση ήταν οικονομικά κίνητρα. Ε, χρηματοδότηση από το κράτος για να αυξηθεί η ε, ζήτηση. Στο παρελθόν είχε γίνει αυτό και είχε βοηθήσει βραχυπρόθεσμα. πρόθεσμα. Η ικανότητα όμως να χρησιμοποιείται αυτό το μέσο είναι περιορισμένη στα περισσότερα κράτη-μέλη λόγω των υπερβολικών χρεών τους ήδη. Αυτό που ήταν η λύση ξαφνικά έγινε πρόβλημα. Ο, οι λόγοι για το πρόβλημα του χρέους είναι διάφοροι στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι επειδή υπήρχαν υπερβολικά πολλές οικονομικές ε, ε δημόσιες δαπάνες σε πολλές οφείλεται στον τραπεζικό τομέα όπου υπήρχαν ε, προβλήματα με τράπεζες που έπρεπε να διασωθούν. Σε άλλες η οικονομική ανάπτυξη ήταν τεχνητή και βασίζονταν σε φυσαλίδες οι οποίες κατέρευσαν με την κρίση και αύξησαν έτσι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Πολλές φορές όμως οφείλεται στο ότι το χρέος αυξήθηκε σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου. Και σε πολλά κρατημέλη έχει ξεπεράσει το 60% του ΑΕΠ. Τα ελλείμματα σε, περίπτωση, σε εποχή ύφεσης δεν ε, δεν εξισορροπήθηκαν από ανάπτυξη και μείωση του χρέους σε άλλες περιόδους. Έτσι, ο συντονισμός ε, για την ασφάλεια και την διακυβέρνηση που υπογράφηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα κυκλικά χρέη εφόσον όμως έχουν μειωθεί τα διαστατικά. Ούτε περιορίζουν τις δημόσιες δαπάνες. Φροντίζουν όμως να μην χρηματοδοτούν αυτές οι δαπάνες από υπερβολική ε, δανειοληψία. <clears throat> Θα πρέπει βέβαια όλοι να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που υπάρχουν στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υποστηρίχθηκε από το λεγόμενο Six Pack. Ταυτόχρονα η εξέλιξη βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να συνοδεύεται από περαιτέρω προσπάθειες να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να εξασφαλιστεί η απασχόληση. Πώς θα γινόταν αυτό ήταν αυτό που απασχόλησε και τα δύο ευρωπαϊκά συμβούλια μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξεμήνου, όπως σας είπα και στο, ε, από το Συμβούλιο του Γενάρη. Προσεγγίσαμε το πρόβλημα από πολλές ε, οπτικές γωνίες. Ελέγχοντας τους προπολογισμούς θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων, εξετάζοντας προσεκτικά τις δαπάνες, ενισχύοντας ε, τους ε, ανέργους, εξετάζοντας τα έσοδα, παραδείγματο χάρη αντιμετωπίζοντας ε, την φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, επενδύοντας στις υπηρεσίες, στις ψηφιακές αγορές, όπως τονίζει μια επιστολή δύο συναδέλφων. Επίσης, ε, ενισχύοντας εκείνους που έχουν χαμηλό εισόδημα, ανοίγοντας ε, πολλούς ε, νέους τομείς, βελτιώνοντας το επιχειρησιακό περιβάλλον και δίνοντας δυνατότητα να υπάρχει μια ψηφιακή διαχείριση, δηλαδή κάνοντας τις σωστές επιλογές για ανάπτυξη και απασχόληση μέσα στα πλαίσια της ε, οικονομικής, ε, του οικονομικού ελέγχου. Ξέρετε ότι το εξάμεινο αυτό είναι ένα ετήσιο μέσο διαχείρισης από τη στιγμή που εκδίδει η Κομισιόν την έκθεσή της μέχρι τη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου που δίνει συστάσεις σε μια κρίσιμη στιγμή. Βέβαια, πολλά από τα μέτρα από την πλευρά της προσφοράς ε, διαρκούν για να έχουν αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά η φορολογική παγίωση έχει πολύ πιο άμεσες ε, επιπτώσεις και αποτελέσματα. Ίσως μπορούμε να αποφύγουμε μια σερίγνωση της, ε, των πιστώσεων και ελπίζω να μπορούν να ε, τύχουν σωστής εκμετάλλευσης τα χρήματα που διαθέτει η, κεντρική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Οι δράσεις της Κεντρικής Τράπεζας και του κυβερνήσεων βοηθούν και είναι πολύ κρίσιμο για τις χώρες να μην διακόψουν τις ε, προσπάθειές τους και να συνεχίσουν με τις προσπάθειές τους. Μέσα στα πλαίσια και της ε, συμφωνίας. Εκτός από την νομισματική αυτή πολιτική, η σφαιρική πολιτική της επαναφοράς της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη μας κάνει να ακολουθήσουμε μια άλλη σειρά μέτρων, ούτω ώστε και από εκεί να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η στρατηγική μας αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο στροφής στην κρίση, παρόλο που βέβαια γνωρίζουμε ακόμα πόσο ευάλωτοι παραμένουμε. Χρειαζόμαστε μία βράχη και μράκρη πρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη. Αυτά αναφέρονται στις στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και τώρα βέβαια και στην πολιτική για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μια πολιτική απασχόληση ιδίω για τους νέους ακόμα και αν η κύρια ευθύνη βρίσκεται στα κράτη-μέλη, μπορεί να δώσει κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το κάνουμε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προσβλέπουμε στην ε, μελλοντική πρόταση δέσμης μέτρων για την απασχόληση της Κομισιόν. Επίσης, για την Ελλάδα χαιρετήσαμε την ε, πρόοδο που επιτέχθη στο νέο ελληνικό πρόγραμμα και έχουμε σαν στόχο να βρεθεί σε βιώσιμο επίπεδο πάλι η ελληνική κυβέρνηση και όσον αφορά την ανεφορία και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα και θα ήθελα να πω σε εκείνου που λένε ότι επιβάλλει τη λιτότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι χώρε της Ευρωζώνης και το ε, Διεθνές Νομισματικό Τομείο προσφέρουν άλλα 130 δις πάνω από εκείνα τα αρχικά 110 δις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις για να μπορεί έτσι να εξασφαλιστεί το 75% των ε, χρεών της προς τράπεζες. Η υποστήριξη της ε, Ένωσης προς την Ελλάδα είναι πάνω από το 100% του ΑΕΠ. Χωρίς αυτή την ε, ενίσχυση θα ήταν πολύ πολύ χειρότερη η κατάσταση της Ελλάδας. Χρειαζόμαστε με την Ελλάδα μια ισχυρή ατζέντα ανάπτυξης τονίζοντας τις προσπάθειες της ε, ε, επενδύσεις και το δυναμικό της Ελλάδας. Θα πρέπει η Κομισιόν να βοηθήσει τεχνικά την Ελλάδα για να πετύχει σε αυτούς τους στόχους. Επίσης η Ευρωζώνη επιβέωσε την δέσμευσή της να εξετάσει ε, το πόσο σωστό είναι αυτά τα όρια που έχουν οριστεί μέσω της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα συμφωνήσαν να επιταχύνουν την πληρωμή των, ε, ε, των κεφαλαίων από το ESF. Επίσης υπήρχαν και πολλά άλλα θέματα που συζητήθηκαν για τη Σερβία. Συμφωνήσαμε να της δώσουμε το καθεστώς της υποψηφίου χώρας γιατί ε, κατέφερε πολλά μετά τις προσπάθειές της όπως που διαφάνει και στο διάλογο μεταξύ Βελγραδίου και Πριστίνα. Ελπίζω να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ούτως ώστε να πληρωθούν τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια για την ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, συνεχίσουν να ενισχύουν την περιφερειακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. Ταυτόχρονα περιμένουν περισσότερο, ε, περισσότερο τακτοποίηση των σχέσεων μεταξύ Πριστίνα και Βελιγραδίου. Όσον αφορά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας στο χώρο του Σέγγεν. Είπαμε να τεθεί αυτό στη μεσία διάταξη του Συμβουλίου για τον Οκτώβριο και να ξεβρεθούν όλα τα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία της διαδικασίας αυτής. Στη Συρία, που αντιμετωπίζει μια φοβερή κατάσταση, έχουμε συγκεντρώσει την προσοχή μας σε τρεις κύριες πτυχές. Ανθρωπιστική πλευρά. Καλούμε να σταματήσει αμέσως η βία κατά των αμάχων και οι παραβάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είπαμε ξεκάθαρα ότι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι θα κληθούν να και θα κατηγορηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κοινοτοποιήσει ε, ανθρωπιστικά κονδύλια. Πολιτικά θέλουμε να αυξήσουμε την πίωση στο καθεστώς ε, στην κυβέρνηση της ε, Συρίας και να προβλεφθούν συμπληρωματικά περιοριστικά μέτρα. Καλήσαμε τον πρόεδρο Ασάτ να παρατηθεί όταν αρχίσει η δημοκρατική διαδικασία, οπότε θα αρχίσουμε και εμείς μια νέα σχέση εταιρική. Διπλωματικά ενισχύουμε την ε, στάση της, ε, του Αραβικού Συνδέσμου. <clears throat> Καλούμε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του Ηνωμένου Εθνών, της Κίνας και της Ρωσίας ιδιαίτερα να συνεργαστούν καταβάλλοντας προσπάθειες να σταματήσει η βία. Μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικά χωρίς εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή ήταν μια άποψη που υποστηρίχθηκε ομόφωνα. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει πολύ πιο ε, κοινή εξωτερική πολιτική από ό,τι πολλοί πιστεύουν. Στις πιο επικίνδυνες περιοχές της Ένωσης του κόσμου, οι 27 εργάζονται χέρι με χέρι. Είναι κάτι που πολλοί φορές παραβλέπετε. Τέλος, είχα την τιμή και 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβούλου να αποφασίσουν να μου ζητήσουν να συνεχίσω για άλλο δύο χρόνια στο αξίωμα μου Προέδρου του Συμβουλίου. Οι 17 μάλιστα του χώρου ε, Βερό μου ζήτησαν να προεδρεύω των συνεδριάσεων κορυφής τη Ευρωζώνης. Δεν θα απορρίσετε που η κύρια μου προτεραιότητα παραμένει η οικονομία. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή οικονομική βάση για να προωθήσουμε το, το κοινωνικό μας πρότυπο, να προωθήσουμε την απασχόληση και για τους νέους και αυτό είναι ο μόνος τρόπος, ο μόνος τρόπος να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή που να είναι ισότιμος με το δυναμικό μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τιμή μου που μπορώ να συνεχίσω την εργασία μου στην τόσο αποτελεσματική αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Φαν Ρομπόη. Το λόγο να μέσα στο Επιτροπή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπερόζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω ήδη συγχαρεί τον πρόεδρο Φαν Ρομπόη για την επανεκλογή του. Θα ήθελα εδώ να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να εκφράσω τη βαθιά εκτίμησή μου για τη δουλειά που έχει επιτελέσει τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Προσδοκώ με πολύ μεγάλη χαρά να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του για να φτιάξουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη που θα εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών και θα είναι ε, ακόμα πιο δυνατή στο διεθνέ στερέωμα. Έχει ήδη υπογραμμίσει ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την έκβαση των ε, συζητήσεων στο Συμβούλιο, ειδικότερα ως προς την κατάσταση διεθνώς στη Συρία, στο Ιράν, αλλά και την παραχώρηση του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας στη Σερβία. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι προχωρά προς περισσότερη σταθερότητα και περισσότερη ανάπτυξη. Λιγότερη ένταση βρίσκεται γύρω από τη ζώνη του ευρώ. Δεν έχουμε βέβαια ξεφύγει από την κρίση. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας με την ε, θέση σε ισχύ των δικλείδων ασφαλείας. Όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας είναι απαραίτητα στοιχεία για μια πιο χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Έχω πει επανειλημμένως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και αλλού ότι δεν θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στην βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης, αλλά και στην ανάπτυξη, την έξυπνη ανάπτυξη, την αηφόρο ανάπτυξη, την συμπεριληπτική ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει όλους. Αυτό είναι κλειδί για το μέλλον και παραμένει βασικός στόχος της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισης μας με τον οδικό χάρτη προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, τον οποίο παρουσίασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτή η προσέγγιση τη χάνει όλο και μεγαλύτερη στήριξη τώρα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση βεβαίω. Παρόλο που μένουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μια συνολική προσέγγιση δηλαδή συμφωνία ε, συνολική για να ανταποκριθούμε στα προβλήματα στην Ελλάδα. Δεύτερον, δημοσιονομική σταθερότητα και ανάπτυξη που θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών και στοχευμένων επενδύσεων. Ας ξεκινήσουμε με την Ελλάδα. Ορισμένοι συνεχίζουν να λένε ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Και ρωτώ γιατί. Γιατί να μην μπορεί η Ελλάδα να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατό, είναι εφικτό. Η ελληνική κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ελληνικό πιστεύουν ότι αυτό είναι δυνατό. Η Συμφωνία για τη Συμμετοχή των Ιδιωτών, το Public Sector Involvement, το PSI και αυτό δείχνει ότι όλοι πιστεύουν ότι αυτό είναι εφικτό και δυνατό. Ε, ο ελληνικός λαός καταβάλει προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Βρισκόμαστε σε στενέ συνομιλίε και συνεργασία με τον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο και την ομάδα του, τους ώστε βασικέ αποφάσει για την ανάπτυξη να ληφθούν αμέσω. Συμφωνήσαμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μα σε συγκεκριμένε προτεραιότητε κλειδιά. Προώθηση ενό περιβάλλοντο πιο φιλικού προ τι επιχειρήσει, παροχή ρευστότητα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, άρση εμποδίων, ούτω ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα διαρθρωτικά ε, τα μία Είναι τομείς αυτή που η Ελλάδα μπορεί να σημειώσει πρόοδο αμέσως, όχι μετά από μήνες ή μετά από χρόνια. Και βεβαίως γίνεται συζήτηση για το πώς θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά ε, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Χθε είχαμε μια συνάντηση με τον διοικητή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εξετάζοντα τρόπου που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Τι επόμενε εβδομάδε, μαζί με τον Αντιπρόεδρο κύριο Όλι Ρεν, θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανακοίνωση για την πρόοδο που έχει ήδη σημειώσει η Ελλάδα, θέτοντα επίση συγκεκριμένου στόχου για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν τον οδικό χάρτη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, ούτω ώστε να εξευρεθούν τελικέ λύσει. Είναι απαραίτητο ο οδικό χάρτη και η δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί χωρί αυτήν δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη των επενδυτών και χωρί εμπιστοσύνη δεν θα υπάρχουν θέσει απασχόληση και ανάπτυξη. Το Συμβούλιο με τα συμπεράσματά του δείχνει τη δέσμευσή του Βέβαια, με το σύμφωνο ε, ε, Europlus Plus, ε, αυτό το σύμφωνο δεν ήταν προτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί προάγει την διακυβερνητική μέθοδο και όχι την κοινοτική μέθοδο. Ωστόσο 25-26 στις 27 χώρες συμμετείχαν, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρώπης και δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναντίστρεπτο. Δεν ε, θα πάμε προς τα πίσω και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους ε, επενδυτές. Η σταθερότητα είναι σημαντική για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τη δέσμη μέτρων, την εξάδα των μέτρων, όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάστασή μας μας βοηθούν να λύσουμε το πρόβλημα έχουν τα συμβαλόμενα μέρη ε, συμφωνήσει να ενσωματώσουν στη δική τους νομοθεσία όλες αυτές τις ρυθμίσεις τα επόμενα πέντε χρόνια. Και έχουμε και την διάδα των μέτρων, τη δέσμη δύο μότρων, ούτω ώστε να υλοποιηθούν ε, τα προβλεπόμενα στην ε, δημοσιονομική συμφωνία. Βεβαίως, η συμφωνία αυτή δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να καλύψει όλα τα οικονομικά στοιχεία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ένωσης. Καλύπτει τα πιο βασικά την εσωτερική αγορά, την κοινωνική και την ε, οικονομική συνοχή. Βεβαίως ε, η ενιαία αγορά και η κοινωνική συνοχή είναι θέματα που θα λύνονται και θα δρομολογούνται καλύτερα βάσει της κοινοτικής μεθόδου. Η υλοποίηση της ατζέντα για την Ευρώπη του 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι ο στόχος μας. Και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη αλλά όχι αρκετή. Έχουμε επανειλημμένως πει ότι βεβαίως χρειαζόμαστε δημοσιονομική σταθερότητα από τη μία και οικονομική ανάπτυξη από την άλλη. Και τα δύο μαζί χρειαζόμαστε. Πολλά στοιχεία αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Ε, η έλλειψη απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η στοχευμένη επένδυση. Βεβαίως και χρειαζόμαστε επενδύσεις και μάλιστα στοχευμένες. Και η αναζωπήρωση του εξωτερικού εμπορίου, του εμπορίου με τις εξωτερικές αγορές. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα για να υλοποιήσουν ε, τις αποφάσεις που έχουν πάρθει και που αποτελούν έκφραση της πολιτικής βούλησης. Υπάρχει απόσταση μεταξύ αυτών και αυτών που γίνονται στην πράξη. Δεν συζητούμε μόνο στις Βρυξέλλε στο κτίριο γίου τους Λήψιου όπου συνεδριάσει το Συμβούλιο. Πρέπει όλα αυτά να μεταφράζονται στην πράξη, στα κράτη, στις περιφέρειες, στις τοπικές κοινωνίες. Και χρειαζόμαστε την προοπτική της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής συμπερίληψης, διότι βεβαίως διαπιστώνεται άνοδος της φτώχειας σε πολλά κράτη-μέλη. Έχω ήδη τονίσει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι πολιτικώς αποδεκτές και κοινωνικώς αποδεκτές από τους πολίτες. Εξού και χρειάζεται κοινωνικές κοινωνικός διάλογος και γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στον τριμερή ε, κοινωνικό διάλογο μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και ε, υπόλοιπης οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει η προσέγγιση να είναι δίκαιη. Τα βάρη και τα ωφέλη να μοιράζονται από όλους και σε όλους. Ο δίκαιος χαρακτήρας ήταν το βασικό κίνητρο ε, πίσω από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φόρο επί των χρηματιστηριακών ε, συναλλαγών. Μια πρόταση που κάναμε πέρσι. Η φορολογία είναι θεμελιώδης συνιστόσα για την ανάκαμψη των οικονομιών μας. Αυτό έχει υποθεί επανειλημμένως και από πολλά Ένα τρεις ευρώ χάνεται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με λόγο φόρο αποφυγής και φόρο διαφυγής. Αν συγκρίνουμε αυτό το 1-3 ευρώ με αυτό το οποίο χρειάζονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί για να είναι ισοσκελισμένοι, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Μια ενιαία αντιμετώπιση, στεναρή αντιμετώπιση από όλου μα θα είναι αρκετή για να λυθεί το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει προτάσει για την καταπολέμηση τη φόροδιαφυγή και φόροαποφυγή Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν λόγο τα κράτη-μέλη να καθυστερούν και να μην υιοθετούν την οδηγία τη σχετική που έχει να κάνει με τις φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες ε, και την οδηγία που έχει να κάνει με το ε, με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις σε θέματα φορολογίες. Μιλώ για αυτό το κενό υλοποίησης το οποίο ε, παρατηρούμε. Δηλαδή τα κράτη-μέλη υιοθετούν θέσεις στο Συμβούλιο και μετά αυτές οι θέσεις δεν υλοποιούνται πρακτικά πίσω στις χώρες, των, στις χώρες τους. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό υλοποίησης μεταξύ της πολιτικής βούλησης που εκφράζεται στο Συμβούλιο και της εφαρμογής στην πράξη μετά ε, τις εκάστοτε πρωτεύουσες. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι ε, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης και χαίρομαι για τη στάση που έχει οθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτησή του ε, με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Χαίρομαι επίσης διότι έγινε δεκτή η πρότασή μας για τα ομόλογα έργων, τα project bonds και έγινε δεκτή και η πρότασή μας για τις δράσεις προτεραιότητας, για την ετήσια αναθεώρηση ε, για την οικονομική μεγένθηση, για την μέτρηση των στόχων που επιτυχάνονται ανάλογα με την τήρηση του προϋπολογισμού. Όλα αυτά θα, οθήσουν, θα βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα βελτιώσουν τη ζωή μας καθημερινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα τέλη Ιανουαρίου έχει αναλάβει δράσεις για να μειωθεί δραστικά η ανεργία των νέων και για να προβλεφθεί στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η απάντηση για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Από το άτυπο Συμβούλιο του Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουμε επισκεφθεί 8 κράτη-μέλη και έχουμε προσπαθήσει να βρούμε τρόπους ώστε περισσότεροι νέοι να εντάσσονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου κάπου εδώ λέγοντα ότι έχουμε διανύσει πραγματικά πραγματικά πολύ μεγάλη απόσταση και έχουμε ε, ε, κάνει άλματα ε, προς την επίλυση των προβλημάτων. Δεν θα πρέπει να δραματοποιούμε την κατάσταση και να μεμψημυρούμε. Θα πρέπει να δουλεύουμε σκληρά για να διατηρήσουμε μια οικονομία της αγοράς με κοινωνικό χαρακτήρα. Το περιβάλλον γύρω μας είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια οικονομία που να προωθεί την ανάπτυξη όντας σταθερή μέσω ανάληψης ευθυνών από όλους μας και μέσω έκφρασης ελληλαγγύης από όλους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για το λεπτά στη του. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καταρχά θέλω να σα συγχαρώ κύριε Βαν για το νέο διορισμό σα και σα εύχομαι ό,τι καλό για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Όλοι έχουμε ανάγκη από σωστέ προτάσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Δύο μαθήματα από την κρίση. Πρώτον, ανάκαμψη των εθνικών οικονομικών στοιχείων. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Η υπογραφή τα τελευταίες πριν από δέκα μέρες είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι μια νέα δέσμευση και υποχρεώνει τους εταίρους, θα έλεγα, να επιδείξουν πνεύμα πειθαρχία και σεβασμού των ανηλυμένων υποχρεώσεων. Περιμένουμε από τα κράτη-μέλη πολλά. Περιμένουμε επίσης πολλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θεματοφύλακα της συνθήκης και οι μεγαλύτερες χώρες έχουν παραβιάσει το σύμφωνο σταθερότητας. Κάποιος πρόεδρος μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε χαρακτηρίσει το σύμφωνο αυτό ανόητο. Νομίζω όμως ότι και το εξαπλό πακέτο και το διπλό πακέτο είναι χρήσιμα μέτρα, αλλά δεν φτάνουν από μόνα τους. Το δεύτερο μάθημα από την κρίση είναι η διαρκής και σε συνέχεια ανάπτυξη που να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Εδώ φοβάμαι ότι από την αρχή της κρίσης δεν έχει γίνει τίποτα. Το Συμβούλιο Κορυφής τον Ιανουάριο αρκέστηκε στο να κάνει κάποιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη χωρίς, θα έλεγα, συντονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ δραστήρια. Αλλά αυτές οι δραστηριότητες θα γινόντουσαν καλύτερα κατανοητές εάν δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης και απασχόλησης. Μου κάνει εντύπωση η δυσκολία με την οποία πάρα πολλές χώρες εφαρμόζουν τους κανόνες για τους οποίους έδωσαν μάχη όμως. Και εδώ περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να βάλει τα κράτη-μέλη στο σωστό δρόμο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει θα έλεγα δύο δρόμους και θα το κάνουμε μάλιστα επίσημα και με μια επιστολή προς την Επιτροπή. Καταρχάς, στο τέλος του χρόνου έχουμε 20 χρόνια να γιορτάσουμε για την ενιαία αγορά. Όμως 20 χρόνια μετά υπάρχουν τουλάχιστον 150 τεράστια εμπόδια για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ όχι μόνο οι κανόνες που αποφασίστηκαν να εφαρμόζονται σωστά, αλλά να προταθεί και ένα νομοθετικό πακέτο με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι επίγον έτσι ώστε έστω και με αργό ρυθμό να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποιους λίγους πόντους ανάπτυξης. Ο τριτογενής τομέας είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία στα οποία υπάρχουν προβλήματα. Και πολλές φορές για τα φάρμακα σαν παράδειγμα Πολλές φορές ε, για παράδειγμα στα φάρμακα οι τιμές κυμαίνονται από το 1 στο 3 για τα φάρμακα. Λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε για να δράσουμε και δεν μπορούμε να τα κάνουμε επίσης και όλα μαζί και γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει με μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία σε 10 τομείς της εσωτερικής αγοράς. Η δεύτερη γραμμή που προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι απαραίτητες επενδύσεις για την πολιτική της ανάπτυξης. Προτείνουμε προς την κατεύθυνση αυτή να κρατήσουμε, ε, να εξασφαλίσουμε ένα τμήμα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων των κρατών μελών αποκλειστικά για θέματα ανάπτυξης αλλά που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε και περισσότερους ιδίους πόρους. Ένα ευρώ το οποίο επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και δημιουργεί 5 ευρώ σε επίπεδο επενδυτικό. Θυμίζω, 4 δις βάλαμε στην ενέργεια το 10 και αυτά γέννησαν σε εισαγωγικά 22 δις επενδύσεις. Λέγω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχουν ανάγκη σήμερα οι συμπολίτε μας είναι η απασχόληση, είναι οι θέσεις εργασίας. Θέλουμε μια, ένα μικρό ρυθμό ανάπτυξης καταρχάς και ένα ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης αργότερα. Το δημοσιονομικό ε, σύμφωνο νομίζω ήταν μια προϋπόθεση. Τώρα όμως θα πρέπει να καταπολεμήσουμε συγκεκριμένα προβλήματα όπως η φοροδιαφυγή. Αναφερθήκατε σε αριθμητικά στοιχεία τρομακτικά υψηλά. Η ολοκλήρωση λοιπόν της εσωτερικής αγοράς και η διάθεση συγκεκριμένων ποσών διασφαλισμένων για την ανάπτυξη στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα δημιουργήσουν αυτές τις θέσεις απασχόλησης που θέλουμε. Ευχαριστώ κύριε Τόλο. Το λόγο για την ε, ομάδα Συλλογιστών και Δημοκρατών ο κύριο Φόποντα, πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καθ' ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο Φανεροπόη για την επανεκλογή του. Θα υπάρχουν πολλέ ε, συζητήσει, πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε. Δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ το Συμβούλιο για την απόφαση του για τη Σερβία. Νομίζω για τη Σερβία, την περιοχή και για το Κωσυφοπέδιο είναι η σωστή απόφαση. Δυστυχώ δεν υπήρχαν θετικέ ε, αποφάσει όσον αφορά το Σένιεν με τη Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι λαοί τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αξίζουν τη διεύρυνση του Σένιεν και ελπίζω να γίνει γρήγορα. Αυτό που με όχαρε ήταν αυτό που είπε ο πρόεδρος Σαρκοζή στο τέλος της ε, συνόδου, ότι ίσως διακοπεί η εφαρμογή του Σέγγεν. Μα τι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε πάλι να χρησιμοποιούμε τα διαβατήρια μας για να έρθουμε στο Στρασβούργο. Δεν μπορεί να ήταν σοβαρό αυτό, κύριε Πρόεδρε. Und wenn, und wenn die Sprecherin von Präsident η εκπρόσωπος του Προέδρου ε, είπε ότι οι σοσιαλιστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρεμποδίζουν την εξέλιξη του Σέγγεν. Όχι, εμείς θέλουμε να πάμε προς τα εμπρός στην Ευρώπη και όχι προς τα πίσω. Καλούμε τον πρόεδρο Σαρκοζή να μην περάσει σε ε, εθνιστικιστικά και αντιευρωπαϊκά ε, μηνύματα. Ας παραμείνουμε ρεαλιστές και ας αναγνωρίσουμε την Ευρώπη, ας δούμε σταθερή προς την Ευρώπη, θα είναι καλό και για τον πρόεδρο Σαρκοζή. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να περάσω τώρα σε οικονομικά θέματα. Σε ένα γερμανικό περιοδικό διάβασα σε μια συντάρρευση πώς θέλετε να διατηρήσετε το σύστημα ζήτησης και ε, προσφοράς εάν δεν ασχοληθείτε με εκείνους που θα πρέπει να αγοράσουν τα προϊόντα αυτό. Θέλουμε ένα σύστημα που να μπορούν εκείνοι με τα χαμηλά οικοδήματα να μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέλιξη. Είναι ε, μία μία δήλωση του Χάρη Μπελαφόντα κανού, όχι πολιτικού οικονομολόγου, ένας ε, ε, τραγουδιστής του κατάλαβε τα πράγματα πολύ καλύτερα από πολλούς οικονομολόγους και πολλούς πολιτικούς. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς να υποστηρίξουμε τη ζήτηση, να υποστηρίξουμε τους οικονομικά αδύναμους. Αλλά πολλές φορές γίνεται το αντίθετο, όπως στην Ελλάδα παραδείγματο χάρη ή και στην Ισπανία. Αυτό που πετυχαίνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Λιγότερη ανάπτυξη, λιγότερη απασχόληση, όχι περισσότερη, λιγότερα έσοδα του κράτους και λιγότερους φόρους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τόσο, τόσο αργά αντιδράσαμε για την ανεργία των νέων. Έχετε δίκιο κύριε Φανιλόπαη. Αντιδράσαμε και το Συμβούλιο Αντέδρασε, αλλά από το 2008 αυξήθηκε σφαιρικά η ανεργία των νέων. Τι θα πούμε στους νέους που δεν βρίσκουν θέση εργασίας. Είναι σκανδαλώδες ότι η νεολαία της Ευρώπης πάει σήμερα στην Αργεντινή, στην Αγγόλα και στη Βραζιλία για να βρει δουλειά. Είναι σκανδαλώδος ότι έχουμε σήμερα νέους που εργάζονται για ένα κομμάτι ψωμί. Τι θα κάνουμε με αυτή τη γενιά των ε, μιλεόρο που λένε στην Ιταλία εικονμένο με μιλεόρο. Πώς θα κερδίσουμε τους νέους αυτούς για την Ευρώπη. Η ομάδα μου θέλει μια εγγύηση για απασχόληση και παιδεία. Έχετε δίκιο ότι αυτό είναι εθνικό έργο. Και οι προπολογισμοί το ίδιο όμως και ασχολείται η Ευρώπη. Η δική μου ομάδα θέλει η Ευρώπη να ασχοληθεί με τους νέους, να τους δώσει μια δυνατότητα εκπαίδευσης ή απασχόλησης. Γιατί αυτό είναι το κοινωνικό πρότυπο Ευρώπη. Και θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα και πιο στο πρόεδρο Τράγκη της ε, Κεντρική Τράπεζα Ίσως παραγνωρίστηκαν αυτό που είπε. Το κοινωνικό πρότυπο Ευρώπη δεν πέθανε. Δεν επιτρέπεται να πεθάνει. Εμεί οι σοσιαλδημοκράτε είμαστε υπέρ του να επιζήσει. Ίσως να πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε, αλλά αυτό είναι τμήμα τη δική μα ταυτότητα που θα προασπίσουμε πάση θυσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντα. Πολλοί νομίζω ότι υπάρχει αντίσταση στι μεταρρυθμίσει μεταξύ των πολιτών. Η αντίσταση αυτή υπάρχει γιατί οι πολίτε βλέπουν ότι δεν υπάρχει δίκαια πολιτική όταν ο πρόεδρος Παρόζο δικαίως αναφέρεται σε μελέτη για την φοροδιαφυγή και βλέπουμε πόσο άδικα είναι τα φορολογικά συστήματα και ότι πολλές φορές ακριβώς οι πλούσιοι δεν πληρώνουν φόρους. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και χαίρομαι με αυτό που είπε ο πρόεδρος Παρόζο και ο κύριος ε, Φων Ρόμπαϊ πολλά βήματα γίνονται μπροστά αλλά δεν αρκούν και θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε μια πιο δίκαια κοινωνικά πολιτική και τότε θα δεχθούν οι πολίτες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αυτό που δεν θέλουν να εγκαταλείψουμε αυτό το κοινωνικό πρότυπο που είναι η Ευρώπη, το κοινωνικό μοντέλο που η Ευρώπη θα προσπίσουμε πάθη σε θυσία όπως σας είπα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Σφόμποτα, υπάρχει μια ερώτηση από τον συνάδελφο Ρούτη. Θέλετε να τη δεχτείτε, παρακαλώ. Κύριε Σβόμποντα, μας δείξατε το διαβατήριό σας. Αναφερθήκατε και στον Νικολά Σαρκοζή μάλιστα. Τον ονοματίσατε. Γνωρίζετε ότι ο Νικολά Σαρκοζή ήταν πάντα υπέρ του Σέγγεν. Γνωρίζετε ότι ο Νικολά Σαρκοζή δεν θέλει να καταργήσει το Σέγγεν, θέλει να το ενισχύσει. Ξέρετε πως ε, είναι ας πούμε τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς ασφάλεια. Γι' αυτό να σας θέσω ένα ερώτημα κύριε Τσέποντα. Ναι ή όχι. Θεωρείτε ότι η ρύθμιση Schengen γίνεται αντικείμενο σωστής διαχείρισης. Καταρχήν κύριε ε, ε, συνάδελφοι, κάθε φορά που βγάζω το διαβατήριό μου θα σκέφτομαι Σαρκοζή, ιδίω αν έχει περάσει στην ε, ε, σύνταξη και δεν ε, είναι πια στην πολιτική. Ασφάλεια και Σέγγεν βέβαια πάνε μαζί. Σας ρωτώ όμως, γιατί εξακολουθεί το Συμβούλιο να παρεμποδίζει και η Ρουμανία και η Βουλγαρία παρόλο που τηρούν τις προϋποθέσεις να μην είναι στο Σέγγεν. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να σας υποβάλω. Γιατί ακριβώς ε, δημιουργήθηκε εκεί η ασφάλεια λόγω των μέτρων που εθετήθηκαν. Και είναι παράνομο που διαδιευρύνουμε το σένκε και σας το λέω αυτό, το να το αμφισβητήσει μέσα στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας που το κάνει ο πρόεδρος ε, Σαρκοζή, αυτό πραγματικά είναι καταδικαστέο, γιατί είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της Ευρώπης στο Σέγγεν και δεν πρέπει να το διαφυσπίσουμε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε, γιατί μας δείχνει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε ελεύθερα τα, ε, τα σύνορα, να μπορούμε να κυκλοφορούμε χωρίς διαβατήρια. Αν δεν το αρέσει του κυρίου ε, Σαρκοζή αυτό είναι δικό του πρόβλημα αλλά εμείς και ο κύριος Ολόντ είμαστε υπέρ της ασφάλειας και της ελευθερίας. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο του ο κύριο Φερχόφσατ έχει το λόγο. Δεν είχα την, πρόταση, την πρόθεση να ανακατευτώ, αλλά κύριε Οντί, να είμαστε σοβαροί. Όταν λέει κάποιο ότι οι μισοί μετανάστε πρέπει να φύγουν από τη Γαλλία, όπω είπε ο πρόεδρο Σαρκοζή, όταν επιτίθεται ταυτοχρόνω στου άλλου εταίρου στη συνθήκη του Σέγγεν ω προ τα προβλεπόμετα εκεί. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ε, ποιο είναι τελικά ο υποψήφιο τη άκρα δεξιά ο Λεπένιος, η Λεπένη ή ο Σαρκοζή. Όταν βλέπω πώς εξελίσσεται σαρκοζη οταν βλεπω πως εκστρατεία στη Γαλλία, πραγματικά εκ, εκπλήσωμαι. Είναι πρωτοφανή τα πράγματα που γίνονται ε, πρόεδρος ε, αυτή τη στιγμή της Γαλλίας ε, να κάνει προεκλογική εκστρατεία και να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκφράσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να επανέλθω στη συζήτηση που κάναμε πριν από την παρέμβαση του κυρίου Οντί. Καταρχάς, να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε και Φαν Ρομπόη. Έρχονται και φεύγουν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και πάντοτε παρατηρούμε εμείς μια φοβερή αυταρέσκεια από την πλευρά τους. Πιστεύετε πραγματικά ότι έχουμε φτάσει στο σημείο καμπή στη κρίση όπου τα πράγματα θα αντιστραφούν προς το καλύτερο. Πιστεύουμε ότι με τις προσπάθειες του κυρίου Μόντι και του κυρίου Ραχώη θα ε, λύσουμε το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θα ε, ξεκαθαρίσει τα πράγματα, το χάος που επικρατεί, ότι αρκεί να συγχωνευτούν τα δύο ε, ε ταμεία διάσωσης με 750 δις ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική έχουν καταλαγιάσει οι αγορές γιατί ο, ο, και ο διοικητής Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζάς αγόρασε χρόνο τυπώνοντας 1-3 ευρώ σε χρήμα. Βλέπουμε λοιπόν τα αποτελέσματα του τυπώματος χρήματος. 1-3 ευρώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτή δεν είναι μια πραγματική λύση, δεν είναι μια διαρθρωτική λύση. Μπορεί να λειτουργήσει για λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες, αλλά δεν είναι οριστική δομική λύση στην κρίση. Και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η δομική επίλυση της κρίσης. Χρειαζόμαστε ε, μερική αμοιβεοποίηση, αν θέλετε, του χρέους. Στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών μας είπαν κάντε το, ε, δημιουργήστε αυτό το Ταμείο Διάσωσης ε, με δομικές διαθροτικές λύσεις, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι έχουν δει το φως παντού αλλού στον κόσμο, εκτός από εμάς. Δηλαδή το χρέος άνω του 60% θα πρέπει να... <coughs> Ε, μοιραστεί έτσι ώστε όλοι να, να πληρώνουν λιγότερα επιτόκια, να είναι πιο βιώσιμα και να έχουμε τη δικλίδα ασφαλείας των 2,3 ε, ε, ευρώ. Αν συγχωνεύσετε αυτά τα ταμεία διάσωσης που έχετε, ουσιαστικά έχετε πυροσβεστήρα, δεν έχετε φραγμό προς την πυρκαγιά που μας απειλεί. Ε, μπορεί να κατασβήνετε να καταλαγιάζετε λίγο τις φλόγες στην ε, Ελλάδα ή στην Ιρλανδία ή στην Πορτογαλία, αλλά δεν μπορείτε ε, να λύσετε το πρόβλημα όταν η φωτιά θα επεκταθεί στην Ιταλία και στην Ισπανία. Δεν, δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται νέα νομοθεσία. Να υιοθετήσουμε νέα νομοθεσία μόνο εάν περιλαμβάνει την γνωστή πρόταση του να έχουμε πραγματικά αυτό το firewall. Αυτά λοιπόν για τη δημοσιονομική κρίση. Για τη Συρία και άλλα σώματα νεκρών γυναικών, παιδιών, μαχαιρωμένων ε, βρέθηκαν στη Χόμς χθες. Και από ό,τι φαίνεται ε, η διεθνής κοινότητα δεν αντιλαμβάνεται πολύ καλά την κατάσταση στη Δαμασκό. Θα πρέπει λοιπόν να, κάνουμε, να περάσουμε στην πράξη, να αποπέμψουμε τους ε, Σύριους πρεσβευτές, να παρεμποδίσουμε τους πολίτες μας, να τους πούμε να μην ταξιδεύουν προς αυτή τη χώρα, να ε, ε, λειτουργήσουμε όπως ο πρόεδρος Ομπάμα, να φτιάξουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους, να, έχουμε, να προσφέρουμε αρρωγή. αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ιδαλλιώς η μοναδική έκβαση είναι η Συρία να μετατραπεί σε μια νέα Στρεμπρένιτσα, σε, ένα νέο, ε, σε μια νέα Ρουάντα, σε ένα νέο Σουδάν. Και εμείς θα έχουμε υπάρξει μάρτυρες άπρακτοι όλων αυτών, εάν δεν τράσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Φεχορστάτ, ο πρόεδρος Ντόλ έχει να σας υποβάλει μια ερώτηση. Όχι, όχι. Θα ήθελα πολύ απλά ε, να μάθω ποια είναι η αντίδραση του φίλου μου Γκί διότι ε, ο πρόεδρος Σαρκοζή δεν έχει στην κυβέρνησή του ε, το εθνικό μέτωπο ενώ στις κάτω χώρες οι δικοί τους κυβέρνηση δεν έχουν ποτέ καταδικάσει τίποτα και κάτι το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο και πολύ πιο λανθάνων αν θέλετε. Ο... Όταν ε, γίνεται λόγος για την Ελλάδα η οποία θα πρέπει να φύγει από το ευρώ, δεν έχω ακούσει ποτέ τον, τον Κίφερ Χόφστατ να επικρίνει αυτή τη θέση. Ευχαριστώ ο κύριος Φερχόφστατ. Ήμουν ο πρώτος που έχει καταδικάσει τη σιωπή της Ολλανδικής κυβέρνησης για το θέμα ε, των διαδικτυακών αυτών τοποθεσιών που αναφέρονται στους πολίτες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, και σας υπενθυμίζω ότι είναι χριστιανοδημοκράτες ενδεχομένως όπως εσείς. Εγώ τηλεφώνησα στον κύριο Ρόιτερ. Δεν ξέρω αν εσείς τηλεφωνήσατε στους ομολόγους σας και θα τα πω και ξεκάθαρα σήμερα το απόγευμα που θα το συζητήσουμε το θέμα. Ε, εγώ θέλω να υπάρξει μια κοινή θέση για την ε, σχετική διαδικτυακή τοποθεσία. Είναι απαράδεκτη η σιωπή της Ολλανδικής κυβέρνησης. Όμως προτιμώ τη σιωπή της Ολλανδικής κυβέρνησης από τις ε, ε κραυγές και τους αλλαλαγμούς του κυρίου Σαρκοζή αυτή τη στιγμή, τους ξενοφοβικούς. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη φιλία. Πολύ ωραία. Ξανάμετω της των Πρασίνων, ο κύριος Κονπέντιτ. Συνάδελφοι, κύριε Φόν δεν ξέρω αν πρέπει να σας συγχαρώ για αυτά τα οποία ακούσαμε. Θα δούμε τα πράγματα, ο χρόνος θα δείξει. Ελπίζω πάντως η δεύτερη περίοδος εντολής σας να είναι καλύτερη από την πρώτη. Θα επανέλθω στο Σέγγεν λίγο και να πω κάτι το σαφές. Η Γερμανία και η Γαλλία είναι απομονωμένες στο Συμβούλιο. Όλες οι χώρες αρνήθηκαν να επανεθνικοποιήσουν τη διαχείριση του Σέγγεν. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε ό,τι για την Ελλάδα αν σταματήσουμε να προκαλούμε με τους Τούρκους με ανόητα ψηφίσματα στα εθνικά κοινοβούλια, ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε μαζί τους να ασφαλίσουν καλύτερα τα σύνορά τους. Τους βαράμε συνέχεια και μετά παραπονιόμαστε γιατί είναι επιθετικοί απέναντί μας. Λοιπόν, ας ε, σκεφτούμε διαφορετικά πώς θα διασφαλίσουμε τα σύνορα με την Ελλάδα, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν πρέπει να λέμε ανοησίες, ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά τα οποία λέμε. Να μιλήσω λίγο για την οικονομική κρίση. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο χρυσούς κανόν ή θα είναι τριπλός κανόν και χρηματοπιστωτικός και περιβαλλοντικός και κοινωνικός. Τότε μόνο έχει νόημα. Εγώ δεν είμαι κατά του χρυσού κανόνα αυτού του, ε, του δημοσιονομικού, συγγνώμη αλλά αν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχους χρυσούς κανόνες περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, τότε δεν θα έχουμε κάνει τίποτα για τις επόμενες γενιές. Πέραν αυτού, αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι ένα πρόγραμμα ανάκαμψης. Ένα ουσιαστικό πρόγραμμα ανάκαμψης όμως. Διαθέσαμε 4.000 δις μέχρι τώρα για να σώσουμε τις τράπεζες. Εγγυήσεις τα ονομάσαμε, επενδύσεις τα ονομάσαμε, πάρα πολλές μορφές ε, χρημάτων. Το σχέδιο Marshall όμως ήταν το 5% του Αμερικανικού ΑΕΠ. 5% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι 800 δις. Τι σχέση έχει με το 4.000. Λοιπόν, 800 ε, ε, δις δεν είναι κάτι το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες χωρών όπως η Ισπανία, η Ελλάδα κτλ δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με μια πολιτική λιτότητας η οποία πνίγει αυτή τη στιγμή τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε σε άλλη κλίμακα αντίδρασης. Έτσι μόνο θα σώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό σε όλους. Θέλουμε λοιπόν δημοσιονομικά μέσα κατάλληλα για να καλυφθεί το πρόβλημα και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσπαθήσουμε να περάσουμε σε δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα μας διασφαλίσουν την ανάπτυξη σεβόμενη και την πράσινη οικονομία. Τώρα για τη φοροδιαφυγή πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Όσο υπάρχει αυτός ο, ο, φορολογικός ανταγωνισμός στην Ευρώπη δεν θα γλιτώσουμε τίποτα. Στην Ιρλανδία έχετε την Apple και το Facebook, στο Λουξεμβούργο έχετε την Google και την Amazon ενώ τα χρήματα τα δίνει η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Οι εταιρείε αυτέ όμω πληρώνουν φόρο στο Λουξεμβούργο και στην Ιρλανδία. Ε, γιατί είναι αθέμητο ο ανταγωνισμό ο φορολογικό. Αν παραμένει η κατάσταση έτσι, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Δεύτερον, αν θέλετε να καταπολεμήσετε τη φοροδιαφυγή είναι απλό να πείτε ότι όλες οι τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είτε είναι ελβετικές είτε ξένες είτε ευρωπαϊκές πρέπει να δηλώνουν το τι καταθέσεις έχουν όλοι οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν ισχύει αυτό για όλους, τότε δεν θα πρέπει να μπορούν να δραστηριοποιούνται οι τράπεζες αυτές. Αυτό δεν έκαναν οι Αμερικανοί με τη UBS στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και είδατε πώς οι, Ευρω... οι ελβετικές τράπεζες προσαρμόστηκαν και έκαναν τις ανακοινώσεις που έπρεπε. Λοιπόν, υποχρεώστε τα πιστοτικά ιδρύματα να δημοσιοποιούν να δημοσιοποιήσουν τις καταθέσεις των Ευρωπαίων. Είναι μια προσωρινή άρση του τραπεζικού απορρίτου, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος έχει τι. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Τώρα για τη Βοσνία, το Βελιγράδι, τη Σερβία μάλλον και το Βελιγράδι δεν συμφωνώ. Πρέπει να βοηθήσουμε και τη Βοσνία. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι του πολέμου είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν σήμερα και αυτοί που ήταν τα θύματα του πολέμου ούτε σκαμνάκι στην αίθουσα της Ευρώπης δεν τους δίνουμε. Εγώ δεν είμαι κατά τη συμφωνία με τη Σερβία, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τη Βοσνία. Και αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συμφωνίας του Ντέιτον δεν πάμε πουθενά. Για τη Συρία. Ο Φερχόστατ έχει δίκιο. Ο πρόεδρος των φιλελευθέρων έχει δίκιο. Ανθρωπιστική διάδρομη. Πρέπει να το κάνουμε, όχι να λέμε τι θα κάνουμε. Ναι στην απομόνωση της Συρίας. Όλες τις επιλογές, ένοπλες ή όχι, θα πρέπει να δούμε πώς θα επιβάλλουμε ας πούμε τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Άμα δεν το δέχεται αυτό ο Ασάντ πώς θα τους επιβάλλουμε. Θα πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για να τους επιβάλλουμε γιατί αλλιώς η σφαγή του λαού της Συρίας είναι καθημερινή και εμείς απλά παρακολουθούμε ένα έργο το οποίο μπροστά μας περνάει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ευχαριστώ κύριε Κονβέντετ. Το λόγο εξ των συντηρητικών. Ο κύριο Κάλαναν. Ε, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανησυχώ όλο και περισσότερο διότι ε, καταλαμβάνει τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους της εξουσίας μια χαρά αυταρέσκεια. Πολλοί νομίζουν ότι τέλειωσε ο πόλεμος κατά της κρίσης. Πολλοί λοιπόν υπενδύσονται ότι η Ευρώπη τα πάει μια χαρά και ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι κάποιες λίγες μεσογειακές χώρες πρέπει λίγο να φτιάξουν τα δημοσιονομικά τους, αλλά η καινούργια συνθήκη θα τα ρυθμίσει όλα αυτά. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Η αδυναμία οικονομική είναι πρόβλημα για όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης και η νέα συνθήκη είναι άσχετη τελικά. Δύο μέλη της ομάδας μου ε, είχαν την εντυμότητα να πούν ότι δεν έχει νόημα να υπογράψουμε αυτή τη συνθήκη. Άλλοι την υπέγραψαν αλλά δεν πιστεύουν ότι ισχύει για τους ιδίους. Η Ισπανία και οι κάτω χώρε είπαν ότι ούτω ή άλλω δεν πρόκειται να τηρήσουν τι διατάξει που υπογράφουν τελικά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει σπαταλήσει πολύ μεγάλη ενέργεια για να υπογράψει μια συνθήκη η οποία δεν θα αλλάξει τίποτα από τη δομή τη κατάσταση και η οποία ε, θα πάρει αποφάσει που θα καταδικάσει τον ελληνικό λαό σε μια γενιά φτώχεια. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τι προοπτικέ μια από τι πιο μακροπρόθεσμε υφέσει στην ιστορία της, στην οικονομική ιστορία τη ανθρωπότητα, μια κατάσταση του βιωτικού επίπεδου ε, των τελευταίων δεκαετιών. Είναι μια λύση ε, με πολύ μεγάλο τίμημα. Χρειάζονται μέτρα ούτω ώστε η Ελλάδα να οργανώσει μια οργανωμένη χρεοκοπία εγκαταλείποντας το ευρώ, υποτιμώντας το νόμισμά της, προκειμένου να διασώσει βραχυπρόθεσμα την οικονομία της, υιοθετώντα παράλληλα μεταρρυθμίσεις για να ανακάμψει μέσω μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, ε, τα οικονομικά των υπολείπων χωρών είναι εξίσου ε, φοβερά. Επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων υπέγραψαν μία επιστολή προς το Συμβούλιο, 12 μάλιστα, ε, για μια επικοδομητική ημερησία διάταξη για την Ευρώπη. Όμως δεν έτυχε θερμής υποδοχής η επιστολή αυτή. Έχει έρθει πλέον η ώρα να σταματήσετε να ε, συμπεριφέρεστε ως Συμβούλιο ως αν να είστε οι αντιπρόσωποι, οι ε, εκπρόσωποι επικοινωνίας της Γαλλίας και της Γερμανίας. Χρειάζεται να εξετάσετε θέματα ουσιαστικά για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συζητήσατε για την απασχόληση και ζητήσατε να ε, συμπεριληφθεί το θέμα της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ημερήσια διάταξη, αλλά μάλλον εννοούνται μόνο των δικών σας χωρών. Σας ευχαριστώ ε, βεβαίω ε, και σας συγχαίρω μάλλον που, για το νέο διορισμό σας βέβαια, παρενθετικά να πω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε μια αποφασιστική απάντηση από το σύνολο από το σώμα της Επιτροπής, όχι μόνο από ένα-δύο επιτρόπους που καταλαβαίνουν τι πραγματικά διακυβεύεται. Η Επιτροπή θα πρέπει να περνάει περισσότερο χρόνο ε, δουλεύοντας πάνω σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και λιγότερο χρόνο ε, δουλεύοντας πάνω σε ανόητα ε, βίντεο και διάφορες άλλες δράσεις ε, ίσονος σημασίας. Πρέπει πραγματικά να καταργήσουμε τους εμπορικούς φραγμούς και να μην τους επανακατευθύνουμε. Ο πρόεδρος Σαρκοσί είπε προσφάτως ότι είναι πάρα πολύ ξένοι στη Γαλλία και εγώ είμαι ξένος στη Γαλλία και πρέπει να πω ότι ε, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να μπορέσω να μην ξανάρθω ποτέ ε, σε αυτό το κοινοβούλιο εδώ στο Στρασβούργο στη Γαλλία. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι θα χαίρονταν ιδιαιτέρως να μην χρειάζεται να έρχονται στη Γαλλία ε, για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλανάν. Υπάρχει μια ερώτηση του βουλευτή Νάτολ. Δέχεστε. μία ερώτηση του βουλευτή Νάτολ. Δέχεστε, κύριε Καλάναν. Ναι. Θα πρέπει να σας συγχαρώ, αγαπητέ συνάδελφοι. Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και πολύ καιρό είναι ότι η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα μόνη της υιοθετώντα τη δραχμή. Ωστόσο αυτή δεν είναι η θέση του, η επίσημη της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών. Συνάδελφοι, συμφωνείτε μαζί μου ή όχι στο ότι Συμφωνείτε μάλλον με τη θέση της ε, κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών ότι χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική ένωση ή η θέση σας είναι τελείως διαφορετική από τη θέση της δικής σας κυβέρνησης. Απάντηση. Χαίρομαι διότι δεν είμαι ο εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Όμως είναι σαφέστατη η κατάσταση. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν αν επιθυμούν να μείνουν στο ευρώ ή όχι. Ε, και συμφωνώ με αυτό. Εγώ βέβαια έχω τη δική μου άποψη, αλλά είναι θέμα δικό τους να το αποφασίσουν αν θέλουν να παραμείνουν ή να φύγουν. Οι ερετοί εκπρόσωποι του ελληνικού λαού θα ε, λάβουν αυτή την απόφαση. Και ε, το λέω αυτό διότι πραγματικά πιστεύω στην αληθινή δημοκρατία ως προς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ο κύριος Μέρφη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Παρόζο, κύριε Φανβάπη, πραγματικά απορώ κάθε φορά που μένετε σοβαροί όταν λέτε ότι αρχίζει να λειτουργεί η στρατηγική μας, όταν μιλάτε για ανάπτυξη που οδηγεί σε απασχόληση, όταν αναφέρετε σε μέτρα τα οποία είναι μια επίθεση κατά του ιδιωτικού επίπεδου της, ε, των πολιτών της Ελλάδας, όταν οδηγούμε μετά το 2011 ε, σε μια νέα ζώνη ευρώ και όταν μιλάτε για τη δημοσιονομικό σύμφωνο που έχει πλήξει τόσους πολλούς ε, πολίτες. Ο Τζορτζ Όρελ είπε ελευθερία είναι να μπορεί να πει κανένας ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα Και θέλω να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια του άρθρου 3 για τη μείωση του χρέους και του άρθρου 4 οδηγούν σε αυστηρή λιτότητα σε όλη την Ευρώπη, 5,7 δις ε, περικοπή στην Ιρλανδία, δεκάδες δισεκατομμυρίων σε όλη την Ευρώπη, 4,5 δις ε, ε, πληρωμή πάνω από το, από το στόκους. Αυτά όλα δεν σημαίνουν ανάπτυξη, σημαίνουν μείωση της, του ρυθμού ανάπτυξης, επιδείνωση όλων των όρων και γι' αυτό η Ιρλανδία φοβάται αυτή τη στιγμή και η κύρια ρήτρα του φόβου αυτού που εκφράζεται που λέει ότι μόνο μια χώρα που θα υπογράψει αυτό το σύμφωνο μόνιμης λιτότητας μπορεί να έχει πρόσβαση στο ταμείο του ESF. Πώς μπορούν όλα αυτά να ενταχθούν στη συνθήκη. Ποιος πρότεινε αυτό τον εκβιασμό. Μπορεί η Ιρλανδική κυβέρνηση να αντιδράσει να μην υποχρεώνει το λαό να ψηφίσει υπέρ της μόνιμης λιτότητας. Επίσης, δεν έχουν επικυρωθεί ακόμα οι συνθήκε που επιτρέπουν την δημιουργία του ESN και γι' αυτό εάν θέλουμε ε, μπορούμε χωρίς την δαμόγκλου αυτό ε, σπάθη πάνω από το κεφάλι μας να υπογράψουμε ή να μην υπογράψουμε ελεύθερα, να αρνηθούμε δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Μερφή. Ο κύριος Φάρατζ έχει το λόγο. Δυόμιση επιπλέον έτη λοιπόν, ίσως ε, μια ανταμοιβή για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Βέβαια τα, ε, δεν τα είπατε πολύ καλά. Είπατε ότι η τελευταία συνάντηση κορυφής ήταν θετική, ότι φτάσαμε στο σημείο όπου τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Ήμουν έτοιμος να σας πιστέψω, αλλά πραγματικά δεν μιλήσατε για τη στάση πληρωμών. Είπατε ότι δεν υπάρχει στάση πληρωμών, ενώ ξέρουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα υπήρξε ένα τεράστιο πιστοτικό συμβάν Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και να αγνοούμε ότι η καταστροφή γύρω μας έχει αρχίσει να επιτελείται. Νομίζω ότι έχετε παρεστήσει σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Εσείς συνεχίζετε να χαίρεστε το δείπνο σας ενώ ο κόσμος αλλάζει ε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, η ανεργία στην Ελλάδα έφτασε σε τεράστια επίπεδα και η κατάσταση χειροτερεύει. Και ξέρετε ότι επίσης 110 ομολογιούχοι Γερμανοί ε, θα προσφύγουν στα δικαστήρια εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Κατά τα άλλα εσείς φυράτε αδιάφορα. Ίσως και αυτό που είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ότι κανένας δεν αποκλεί να υπάρξει μια τρίτη προσπάθεια διάσωσης της Ελλάδας. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, έχουμε καταντήσει να ζούμε μια φάρσα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Τα κάνουμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Όχι, σταυρώνουμε την Ελλάδα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι για να στηρίξουμε μια προσπάθεια αποτυχημένη. Γιατί ξέρετε ότι άμα πέσει η Ελλάδα θα πέσουν και άλλοι. Όταν οι ηγέτες μας λέγουν εδώ ότι κάποιες πολιτικές αποφάσεις είναι ε, θα έλεγα αναπόδραστες, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όλα αλλάζουν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκόλνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω καταρχάς τον κύριο Σβόμποντα ε, ε, για κάτι. Να του πω ότι από τότε που υπάρχει η συμφωνία του Σέγγεν, εγώ πρέπει να δείχνω το διαβατήριό μου όχι μόνο στα σύνορα, αλλά και στις εσωτερικές ε, μεταφορές. Από το Στρασβούργο στη Λιόν, ας πούμε, πρέπει να δείξω το διαβατήριό μου τη στιγμή που πάω να μπω στο τρένο. Περίεργο είναι. Από τότε που δεν υπάρχει έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα, υπάρχει εσωτερικός έλεγχος παντού. Μυστήριο πράγμα. Δεύτερο, ο κ. Φερχόφσταρτ είναι ένας μεγάλος δημοκράτης, πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία απαγόρευσε ε, το Βλάμς Μπλοκ, την βασική μονάδα της αντιπολίτευσης και που θέλει να απαγορεύσει και το διαδίκτυο και θεωρεί ότι είναι ρατσιστικό να υποχρεώνονται οι άνθρωποι στη Γαλλία να τρώνε κρέατα ασφαγιαστέντα σύμφωνα με το τυπικό του Ισλάμ ενώ δεν είναι μουσουλμάνοι και την ίδια ώρα καίγονται τζαμιά στις ε, Βρυξέλλες. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς ε, ε, ξέρω ότι η αίσθηση που έχετε για την δημοκρατία, η φιλελεύθερη αυτή αίσθηση είναι λίγο περίεργη. Αυτό το οποίο μας απασχολεί σήμερα το ονομάζουμε την τελευταία ευκαιρία. Θυσιάσαμε την Ελλάδα και υποτίθεται ότι προς το παρόν οι αγορές έχουν καθυσυχάσει. είναι ήρεμες. Και μιλάμε τώρα για, ένα, για μια φάση σταθερότητας. Σταθερότητας αρνούμενη τη δημοκρατία βέβαια. Ο συντονισμός του Συμβουλίου είναι συντονισμός που οδηγεί στην προσωρινότητα των θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα έχουμε ένα μείγμα πλουτοκρατίας και έλλειψης ελευθερίας που ε, στην ουσία επιβάλλεται μέσω των αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυταρχικό τρόπο, σκληρά αυταρχικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. ολόκληρου του ΕΛΚ, ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. με κύριε Πρόεδρε Σούλτ, κύριε Πρόεδρε Φένροπα, κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο. Σωστό είναι αυτό που ελέγχθη, ότι δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε. Είναι επίση σωστό όμω και πρέπει να το πούμε ότι ένα τμήμα του έργου μα επιλύεται και ότι βρίσκουμε σωστή άγουσα. Αν θέλουμε να λύσουμε μεγάλα προβλήματα θα πρέπει να ενθαρρυνθούμε από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να δούμε ποια είναι η σωστή και ποια είναι η μεθασμένη άγουσα. Από την άλλη μεριά, αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε του νέου για το μέλλον και για την Ευρώπη, αυτέ οι συζητήσει που είχαμε στην αρχή, προεκλογή εξαρτία ε, τύπου δηλαδή, δεν ωφελούσε τίποτα. Σφάλουν. Όσον αφορά την ανάπτυξη και σταθερότητα. Ναι, θέλουμε μια οικονομικά σωστή εξέλιξη στην Ευρώπη, ούτως ώστε οι άνθρωποι, οι νέοι ιδίω να έχουν μέλλον, θα πρέπει να χειριζόμαστε σωστά τα χρήματά μας. Και αυτό που έγινε πολλές φορές ε, στο παρελθόν να μπορούμε να το ελέγχουμε. Προσεκτικά δηλαδή να ελέγχουμε τα χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξοικονομούμε μέχρι τελευταία πτώση, αλλά ότι διαχειριζόμαστε σωστά. Όλοι κάναμε σφάλματα. Άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λιγότερο. Και ούτε ελέγχαμε σωστά όταν υπήρχαν κάποια προβλήματα. Και αν θέλουμε να οργανώσουμε την ανάπτυξη, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα χρήματα και άλλα προγράμματα και κάτι παραπάνω. Κανεί δεν κατάλαβα τίποτα. Θα σημαίνει να έχουμε τι σωστέ δομέ, τα σωστά κίνητρα. Υπάρχουν κράτη-μέλη και εθνικές οικονομίες που προχωρούν σωστά. Γιατί, γιατί υπήρξαν διαστατικές αλλαγές, γιατί ε, βασίστηκαν στην οικονομία, γιατί και στις επιχειρήσεις, γιατί θέλησαν να μην διακανονίσουν μέχρι το τελευταίο κόμμα οτιδήποτε. Εάν λοιπόν σκεφτόμαστε περισσότερο πού μπορεί να υπάρχει καινοτομία και έρευνα που θα μας προωθήσουν. Θα κάνουμε πολύ περισσότερο για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά οποιασδήποτε δηλώσει, παρά οποιασδήποτε δηλώσεις που κάνουμε εδώ. Χρειαζόμαστε τόλμη, δέσμευση, εμπιστοσύνη στους νέους και γενικά στους πολίτες, λιγότερες διατάξεις, περισσότερη καινοτομία, περισσότερα έρευνα, αλλά όχι μόνο με λόγια, αλλά στην πραγματική πολιτική. Κάθε μέρα που παίρνουμε μια απόφαση. Αυτό θα ήθελα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί ο αριθμός των συνόδων κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων γιατί δεν χρησιμεύουν και σε πολλά πράγματα. Εάν η Ευρώπη τα πάει κάπως καλύτερα, αυτό το οφείλουμε στη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του διοικητή της κύριου Μάριου Ντράγκη. Αντιθέτως, οι, οι συνόδοι κορυφής πάντοτε έρχονται ε, μετά τις εξελίξεις. Ε, και εκφράζουν γενικολογίες για παράδειγμα για την ανεργία των νέων και όλα αυτά τα ευχολόγια εξατμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Σαρκοζή θέλει να ηγηθεί της Ευρώπης και καυχήθηκε ότι ήταν ο πρωτεργάτης της συνθήκης της Λισαβόνας. Ως υποψήφιος τώρα απειλεί να εγκαταλείψει η χώρα του το Σέγγεν. Αλλά δεν έχει αντιληφθεί βεβαίω ότι η συμφωνία Σέγγεν είναι αναπόσπαστο μέρος της συνθήκης στο άρθρο 67 επιβάλλεται, παραθέτω, η απουσία ελέγχου των ατόμων στα εσωτερικά σύνορα. Τέλος της παράθεσης. Επομένως, για να εγκαταλείψει το Σέγγεν, η Γαλλία θα πρέπει να εγκαταλείψει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, τι θέλει να ελέγξει ο πρόεδρος ε, Σαρκοζή τα, ε, τις τόσες πολλές μετακινήσεις στα εσωτερικά σύνορα τα εκατομμύρια τουριστών που σειραίουν στη Γαλλία το καλοκαίρι, τα δύο εκατομμύρια Γάλλων οι οποίοι ε, μένουν σε γαλλικό έδαφος αλλά εργάζονται από την άλλη πλευρά των συνόρων στις γειτονικές χώρες. Όλες αυτές οι λαϊκιστικές εκφράσεις το μόνο που κάνουν είναι να καλύπτουν την ανικανότητα των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι δεν δίνανται να ε, χαράξουν πολιτική ανάπτυξη. Και το είδαμε και με την Ελλάδα όπου επιβλήθηκαν μέτρα που σαν σε κατάρρευσε της εσωτερικής στήριξης, εσωτερικής ζήτησης που οδήγησαν στην χρεοκοπία χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη δραστική περικοπή της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων και στην ε, φτώχεια τους γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο ε, κύριος Λάμστορφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε μια ε, πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη, έτσι λέγεται. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι πετύχαμε με αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο. Δεν πρόκειται για μια στροφή, δεν πρόκειται για τη λύση, δεν πρόκειται για πανάκια. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Από την άλλη μεριά είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός χρειάζομαι ισορροπημένους προπολογισμού με ελάχιστο ε, έλλειμμα αν ε, είναι, δεν γίνεται δυνατόν τίποτα άλλο θέλουμε τροχοπέδι στην Ευρωζώνη για το χρεό θέλουμε την εξάλληψη των παλιών χρεών και δήλωση στις Βρυξέλλες πριν την δημιουργία νέων χρονών θέλουμε το σύμφωνο να κοινοποιείται πολύ πιο γλυγόρα και μόνο οι χώρε οι οποίε προσπαθούν στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο με το λεγόμενο Tupac προσπαθούμε να εξαλείψουμε το χρέος, πράγμα που ε, συμφωνεί η ομάδα μου με αυτό. 16 ως 18 δισεκατομμυρία διαθέτουν τα ζωτικά ταμεία για την Ελλάδα και θα πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Αυτό που έκανε η Τρόικα μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν αρκεί για να κοινοτοποιήσει η ανάπτυξη. Από την άλλη μεριά έχουμε μια συζήτηση σήμερα με εκπλήτη και στην ε, Γερμανία στη Βουλή που οι Δημοκράτες λένε ότι δεν θέλουν να συνυπογράψουν το δημοσιονομικό σύστημα ε, σύμφωνα εκτός αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φόρος που μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι ένα σφάλμα. Θα πρέπει και οι Δημοκράτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την πολιτική σταθερότητα χωρίς να παίζουν αυτά τα κομματικά παιχνιδάκια είναι σημαντικό να προχωρήσουμε επιτέλου όσον αφορά τον έλεγχο σταθερότητα, κύριε και κύριοι. Τελώντα, θέλω να σα χαρώ κύριε Φανελόπη, εσεί, από ό,τι λένε όλοι εργάζεστε πάρα πολύ καλά, παρόλο θεωρώ ότι η θέση σα, όπως υπάρχει στις συνθήκε τηλεφώνε, δεν είναι σωστή. Εμεί θα ήθελα έναν πρόεδρο στην Ευρώπη που να εκλέγεται και άμεσα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο των Πρεσίνων, ο κύριο Καμφέ έχει το λόγο. Ναι, κύριε Μπαρόζο. Έχετε μιλήσει για την φοροδιαφυγή και δικαίω. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μάχη για μας, μια μάχη που έχει να κάνει με την κοινωνική δικαιοσύνη και με την ε, αποτελεσματικότητα των ε, οικονομικών του κράτους. Καλά είναι τα λόγια, ακόμα καλύτερες οι πράξεις. Ποια πίεση ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς βοηθά την Ελλάδα να ανακτήσει τα 100 και 200 δις ευρώ ή και παραπάνω που βρίσκονται στην Ελβετία βάσει εκτιμήσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Βεβαίως η Ελλάδα έχει μεγάλη ευθύνη ε, λόγω της ανικανότητά της πραγματικά να εισπράξει ε, τα βεβαιωθέντα. Όμως, ε, ποια πίεση ασκείται στην Ελβετία για να επιστρέψουν τα χρήματα στην Ελλάδα και να φορολογηθούν. Ο Ντανιέλ Κονμπεντίτ μίλησε για το τι έκανε ο Ομπάμα ε, σε σχέση με την προσωρινή άρση του τραπεζικού απορρίτου ελβετικών τραπεζών. Πού είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξοεδαφικό νόμο, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Πού, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Έχουμε μία, δύο, τρεις χώρες ε, στη λίστα του ΩΣΑ και μετά ε, τίποτα άλλο δεν γίνεται. Ε, δηλαδή ο κατάλογος με τις ε, ύποπτες χώρες ουσιαστικά είναι κενός. Καλές είναι μεγάλες δηλώσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα καλύτερες είναι όμως οι συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις άσκησης πίεσης. Άσκηση πίεση προ τα κράτη-μέλη και σα χρειαζόμαστε εσά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πιέσουμε τα κράτη-μέλη. Και μία τελευταία ερώτηση, όχι για του φορολογικού παραδείσου, αλλά για τη λιτότητα. Στι ανεπίσημε συζητήσει με τι υπηρεσίε σα μα λένε οι εξιομετούχοι σα ότι εάν βάλουμε όλε μαζί τις πολιτικέ λιτότητας, ε, ε, Εάν τις εντάξουμε στο ίδιο οικονομικό μοντέλο και το εξετάσουμε, ουσιαστικά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι πράγματι έτσι ανοίγεται δρόμος για τη μείωση του ελλείμματος. Γιατί μειώνεται τόσο η ανάπτυξη, μειώνονται τόσο πολύ τα δημόσια έσοδα που τελικά καταλήγουμε σε περισσότερο έλλειμμα και όχι σε λιγότερο έλλειμμα. Αυτό έχει φανεί στην Ισπανία, μάλλον θα φανεί στην Ολλανδία και στη Γαλλία ούτω ή άλλω. Η αλήθεια είναι ότι εάν εξετάσουμε τα στοιχεία βάσει τη οικονομική θεωρία, δεν δουλεύει το μοντέλο αυτό. Πότε θα αλλάξετε λοιπόν μοντέλο. Ευχαριστώ. Πριν λίγες μέρες σε μια ελληνική εφημερίδα ήταν, υπήρξε μια γελιογραφία. Ήταν η κυρία Μέρκελ η οποία βαστούσε ένα μεγάλο σταυρό. Και αυτό θα έλεγα είναι κάτι το απαράδεκτο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα ολοκλήρωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει και επιτίθενται η μία στην άλλη, είναι εχθρικές η μία απέναντι στην άλλη και γενικά τα μέτρα τα οποία παίρνετε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση εσείς στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Φυσικά είναι απαραίτητη η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά θα έλεγα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αποφύγουμε την περαιτέρω πολιτικοποίηση των οικονομικών θεμάτων, έτσι ώστε να χαμηλώσουν οι εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Η χώρα μου δεν υπέγραψε το δημοσιονομικό σύμφωνο. Θα υποβάλει τις, το περιεχόμενο του συμφώνου αυτού όπως και άλλα θέματα σε δημοψήφισμα και γι' αυτό είναι απαραίτητο οι πολίτες της χώρας μου να αποφασίσουν μόνοι τους. Ευχαριστώ κύριε Σχούντι. κύριε Μπαρόζο, κύριε Ρομπάη που είστε εδώ απέναντί μου. Πριν δύο χρόνια η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό έβαλαν το λαό της πατρίδας μου σε ένα τεράστιο πείραμα. η ελλάδα αποτέλεσε το όχημα του διεθνούς νομισματικού ταμείου στην ευρωζώνη. σήμερα το διεθνές νομισματικό ταμείο είναι κατά θεσμικό τρόπο στην ευρωπαϊκή ένωση. το ελληνικό πείραμα μείωση μισθών μείωση συντάξεων μείωση επιδομάτων μείωση δαπανών για τα σχολεία για τα νοσοκομεία κόψιμο των επιδομάτων κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. τα αποτελέσματα. 7% ύφεση πέρσι ένα εκατομμύριο άνεργοι επισήμως ενάμιση ανεπισήμως. κλείνουν καταστήματα εργαζόμενοι δεν πληρώνονται ένας λαό προσβεβλημένος και δυστυχισμένος. χρεοκόπησε η ελλάδα σε βάρος του λαού της σε βάρος της νεολαίας σε βάρος των οικογενειών για να κερδίζουν οι τράπεζες. και τώρα κύριε μπαρόζο κύριε ρομπάι τι αποφασίσατε στο συμβούλιο που συζητάμε σήμερα. αποφασίσατε τη χρεοκοπία της ε- ιδέας της ευρώπης. αποφασίσατε τη χρεοκοπία της ιδέας της αλληλεγγύης. αποφασίσατε να φτιάξετε μια ευρώπη της σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχίας μια γερμανική ευρώπη. αποφασίσατε να φτιάξετε μια ευρώπη που ο ένας θα καρφώνει τον άλλο μια ευρώπη φοβική στους λαούς της μια ευρώπη φοβική στα δημοψηφίσματα και στη φωνή των λαών της. αλλά κύριε μπαρόζο και κύριε ρομπάι οι λαοί δεν χρεοκόπησαν και γρήγορα θα δώσουν απάντηση και θα στείλουν στα σκουπίδια τέτοιες συμβάσεις τέτοια μνημόνια τέτοιες συνθήκες. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. <clears throat> Äh, ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα το πρωί πάρα πολλέ κριτικέ για τι δηλώσει, τι οποίε έκανε ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία για το Σέγγεν. Νομίζω ότι η κριτική που ακούστηκε ήταν λαϊκιστικού τύπου. Βέβαια θεμητό είναι και αυτό. Θα ήθελα να υποβάλω όμως την ίδια ανάλυση αυτό το οποίο υπάρχει στην πρώτη σελίδα όλων των ευρωπαϊκών εφημερίδων κάποιες σημαντικές θέσεις τις οποίες ε, εξέφασε ένας πολύ γνωστός ε, φιλόσοφος, ο κύριος Χάμπερμας ο οποίος θεωρεί ότι το, το δημοσιονομικό σύμφωνο λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή ουσιαστικά αυτού του συμφώνου γιατί δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη αν δεν υπάρξει ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη της δημοκρατίας και μέσα από τα δημοψηφίσματα θα έλεγα εγώ, τότε μόνο μπορούμε να περάσουμε σε αποφάσεις οι οποίες να έχουν αξία. Και θεωρεί ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά θύμα των κερδοσκόπων και λειτουργεί θα έλεγα αφαίρετα απέναντι στους πολίτες της. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Χάμπερ μας, οι αποφάσεις τις οποίες έχετε πάρει είναι λανθασμένες, είναι εις βάρος των λαών, ίσως τις επιβάλλουν τις, επιφάσεις, τις αποφάσεις αυτές οι Λέσχες Μπίλντεμπεργκ, η Τριμερής Επιτροπή και αυτά όλα φύγουν φυσικά και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή της Βετανικής Κυβέρνησης για θέματα ασφαλείας εξέτασε το σενάριο διάλυσης της Ευρωζώνης και το τι θα δημιουργούσε αυτό σε, πολυ, επίπεδο πολιτικής σταθερότητας και τεράστια κύματα προσφύγων που θα έφευγαν από το χάος της Ευρωζώνης και θα ερχόντουσαν στη δική μας χώρα. Είναι σημαντικό το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε μπροστά μας και ακούσαμε αυτή την εβδομάδα ότι ο κύριος Σαρκοζή απειλεί να αποσύρει την Γαλλία από τη συμφωνία του Σέγγεν. Ίσως μεσοπρόθεσμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι σε θέση να διασφαλίσουν την άμυνά τους ε, υπονομεύοντας την ασφάλεια γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι βλέπει ο κόσμος το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Κύριος Μάουρο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κύριος Βόμποντα σχετικά με το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας. Εγώ ίσως δεν πιστεύω με τον ίδιο τρόπο αυτά που είπε ότι οι αποφάσεις του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να αναγνωστούν με ιδεολογικό τρόπο. Είμαστε 500 εκατομμύρια. Ε, τα 75 εκατομμύρια είναι κάτω των 25 ετών. Ε, ενώ βλέπουμε ότι στην Αίγυπτο μόνο τα 60 εκατομμύρια είναι κάτω των 25 ετών. Σε μία χώρα μόνο εννοώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να καλύψουμε με κάποιο τρόπο τα προβλήματα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε τεράστια προβλήματα και βλέπουμε ότι οι ηγετικές τάξεις από τη μία στρέφονται προς κάποιες ειρήνες λαϊκιστικές οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα θέλουν να λύσουν αλλά και από την άλλη προσπαθούν να βρουν λύσεις πραγματιστικές οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να κωδικοποιήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο την ανάκαμψη την οικονομική. Πρέπει λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παράγον που μπορεί να επηρεάσει τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών, μπορεί να τροφοδοτήσει τον δημόσιο διάλογο έτσι ώστε να πιστέψει ξανά στην Ευρώπη. Πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη φάση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι το στρατηγικό μέσο για την ενίσχυση αυτή. Γιατί αλλιώς στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων ανάμεσα σε κυβερνήσεις οι οποίες άγονται και φέρονται από την κοινή τους γνώμη και επηρεάζονται και καταλήγουν σε λαϊκιστικά μέτρα δεν θα πάμε πουθενά. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα από τη Ομάδα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον τον Πρόεδρο της ε, Κομισιόν ότι δεν θα λειτουργήσει το δεύτερο δέσμη για την Ελλάδα όπως δεν λειτουργήσε η πρώτη. Γιατί αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ε, πραγματοποιήσει τις ε, πληρωμές της χώρα αυτή. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο επίσης δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα που οδηγείται έτσι περισσότερο στην ύφεση και μπορεί ακόμη λιγότερο να πληρώσει τα χρέη της γιατί δεν αυξάνεται με τη λιτότητα η ανταγωνιστικότητα της χώρας ούτε η εσωτερική ζήτηση. Το επόμενο και τα επόμενα πέντε χρόνια φαντάζομαι η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ύφεση το 2011 μειώθηκε το ΕΠ κατά 7% και χιλιάδες επιχειρήσεων έκλεισαν. 23% του πληθυσμού είναι άνεργος και δεν δημιουργούνται πια θέσεις απασχόλησης. Το μέσο εισόδημα μειώθηκε κατά 50% από τότε που δρά η Τρόικα. Πού θα δημιουργηθεί ο δυναμισμός για την επιστροφή των χρεών που εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα. Και η δεύτερη δέσμη μέτρων προβλέπει ένα πλεόνασμα 4,5% για πλεόνασμα 4,5% για να μπορούν να επιστραφούν τα χρέη. Πού είναι αυτό όμως. Στη δεύτερη δεσμή προβλέπεται περαιτέρω μείωση των μισθών κατά 25% και 35% μόλις από τους νέους. Αυτή είναι η αλλαγή στην οποία οδηγούμεθα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτης ανάγκης για άλλη μια φορά. Θα πρέπει να ε, βγούμε από το εθνικό αυτό χρέος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί κατά τα άλλα ε, έχουμε μία μεταστροφή αλλά προς το γκρεμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Κατσίν έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε Ρομπάι, αγαπητέ κύριε Μπαρόσο, Χαίρομαι ιδιαίτερως με την απόφαση του Συμβουλίου να παραχωρήσει στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς τα εμπρός και αναγνωρίζει τις ε, μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ε, της Σερβίας. Είναι σημαντικό βήμα για όλες τις γειτονικές χώρες, για τη γενικότερη περιφέρεια και είναι και μια κλίση μια τελευταία κλίση και δραματική κλίση αφύπνισης προς την Μακεδονία, η οποία ματέως περιμένει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης τα τελευταία 7 χρόνια. Παρά τις καθυστερήσεις, ε, παρά τις υποχωρήσεις, το Βελιγράδι έχει αναλάβει τις ευθύνες του και έχει ξεκινήσει ένα σοβαρό διάλογο με την Πρίστινα. Η εφαρμογή όλων των συμφωνιών έχει ξεκινήσει και ελπίζω ότι οι αρχές θα στηριχθούν πάνω σε αυτό την, ε, σε αυτό το δυναμικό το θετικό και θα συνεχίσουν με την καλή την πίστη εφαρμογή της ε, Συμφωνίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Το εκρεμές ε, ζήτημα στη Σερβία σήμερα είναι η συστημική διαφορά και η επιρροή που ασκεί η πολιτική εξουσία προς τη δικαστική εξουσία. Θα πρέπει οι Σέρβοι ηγέτες να κάνουν, καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να επικρατήσει πραγματικά το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή. Και χρειάζονται να κάνουν το παν για να ανοίξουν εγκαίρες στα κεφάλαια 23 και 24 των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω ότι θα διατηρηθεί το φιλόδοξο πνεύμα της ε, Σερβίας ε, στις διαπραγματεύσεις και είναι θεμελιώδου σημασία στο Βελιγράδι να συνεχίσει την επικοδομητική του προσέγγιση προς το κοσφοπέδιο κατά τη διάρκεια και μετά της προεκλογικής εξαρτίας οι παράλληλες δομές στο Βόρειο Κόσοβο θα πρέπει προσεκτικά να αρχίσουν να έρονται έτσι ώστε να εκτελέσουν την εντολή που τους αναλογεί η Γιούλεξ και η ΚΕΦΟΡ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το Μάιο του 2010 έχουν λάβει χώρα πάρα πολλές σύνοδοι κορυφής παράλληλα με πολύ έντονε δημόσιε διαμαρτυρίε των λαών για την απώλεια θέσεων απασχόληση και για τι περικοπές και τη λιτότητα. Οι ηγέτε επικεντρώνονται στη μείωση των ε, ε, δαπανών μόνο. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η κρίση. Για να την αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ριζικά τις απόψεις μας. Η περίοδος κρίσης είναι μια περίοδος άντλησης διδαγμάτων, ούτως ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα παλιά λάθη. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή οικονομία να εξοπλιστεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει τις, τις μελλοντικές προκλήσεις, να επενδύσει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, να δημιουργούνται αηφόρες, βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, να προστατεύεται το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ε, ανάκαμψη των δημοσιονομικών αλλά και για την ανάκαμψη του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή το τίμημα το πληρώνουν οι περισσότερο ευπαθείς, αυτοί που φέρουν τις λιγότερες ευθύνες για την κατηγορία παγίδα που έχει πλήξει την οικονομία. Είναι απαράδεκτο οι νέοι να αισθάνονται αποκλεισμένοι και απορριπταίοι και να μην τους ενθαρρύνουμε να διαδραματίζουν το ρόλο που τους αναλογεί στην οικοδόμηση της Ευρώπης που ονειρευόμαστε. Χρειάζομαστε περισσότερη αλληλεγγύη με όλους τους λαούς της Ευρώπης. Ε, στην εκλογική μου περιφέρεια ε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ούτως ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά προγράμματα επένδυσης σε θέσεις απασχόλησης, σε ανθρώπους, σε υποδομές για να έχουμε πραγματική οικονομική ανάκαμψη. Ευχαριστώ. οι ηγέτες κάνουν ασφαλμένη διάγνωση της ε, ε, κρίσης, λέει ο κύριος Έπινγκ. φτηνό χρήμα οδήγησε σε χρέος και σε φούσκα. Πέρσι ο κύριος Φαν Ρομπάι είπε ότι οι πυλώνες του ευρώ είναι ε, σταθεροί και ισχυροί. Όμως έχει δημιουργηθεί ένα κενό ανταγωνιστικότητας μέσα στην ίδια την ζώνη του ευρώ. Ένα χάσμα μάλλον ανταγωνιστικότητας. Ε, λεγόταν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πάνε καλά. Ενώ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ένεση ενός 3 ευρώ για να μην καταρρεύσουν οι Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Την περασμένη εβδομάδα λέγατε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Ενώ προχθές ο Υπουργό Σόιμπλε είπε ότι μπορεί να χρειαστεί και τρίτο πακέτο διάσωση η Ελλάδα. Ο διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν αναλάβει τα καθήκοντά του προέβλεψε περισσότερη οικονομική ε, συστολή και περιστολή των δαπανών ε, και άλλες χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, ε, κάνουν ένα τεράστιο αγώνα για τα δημοσιονομικά τους. γνωρίζετε ότι δεν σας πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, πρόεδρε Φαν όταν τη μία λέτε τα μεν και την άλλη τα δε. Η κυρία Τζούμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οδηγούν στη θεσμοθέτηση, επίσημη θεσμοθέτηση πολιτικών που έχουν οδηγήσει σε τεράστιες κοινωνικές αδικίες, αν εκτόξευση της ανεργίας, ουσιαστικά τέλος του κράτους ε, πρόνοιας και πίσω από τους ε, όρους αυτούς περί δημοσιονομικής σταθερότητας ουσιαστικά κρύβεται η προσπάθεια καταδίκασης των οικογενειών στην ε, ανεργία και στην απελπισία. Όλα αυτά τα σύμφωνα και οι συνθήκες που έχετε ε, συμφωνήσει και υπογράψει οδηγούν σε απολύσεις, σε ιδιωτικοποιήσεις, ε, σε απαλωτρίωση του εθνικού πλούτου που ανήκει στους λαούς. Ταυτοχρόνως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δίνει τρεις ε, σε ρευστότητα για τις ιδιωτικές ε, τράπεζες. Η υπογραφή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, πέρα από την κοινοτική μέθοδο, ουσιαστικά απειλεί εθνικά κυρίαρχες χώρες ε, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις που τις αφορούν. Είναι μια απικιοκρατικού τύπου αντίληψη υπέρ των μεγάλων δυνάμεων όπως η Γερμανία. Ο Ευρωπαίος εργαζόμενος ε, πραγματικά ε, κάνει ένα τεράστιο αγώνα. Οι Πορτογάλοι εργαζόμενοι θα απεργήσουν προκειμένου να, εκφράσουν την αντίθεσή τους προς όλα αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Ρολάντας Πάξας. Τον Μάρτιο νομίζω ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου βοήθησαν την Ελλάδα τουλάχιστον προσωρινά. Θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε και τις ανάγκες στο μέλλον και να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία μας είπε ο Πρωθυπουργός Μόντι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας ότι για να αναπτυχθεί η οικονομία απαιτείται να υπάρξει και δημοκρατική συνεργασία. Εμείς ακριβώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε σαν υπεύθυνε χώρες να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Οι κυβερνήσεις μας θα πρέπει να εφαρμόσουν υπεύθυνε πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι το α και το ω ε, της ε, οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σεβαστούμε στις αρχές τις οποίες ε, περιλαμβάνει το σύμφωνο το δημοσιονομικό. Αν σεβαστούμε την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη, τότε θα μπορέσουμε να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνον τότε. Ευχαριστώ. Κύριε Πάξας. Κλάες, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης και της 2ης Μαρτίου στο σημείο 44 για να είμαι επακριβέστερος λέγουν τα εξής. Λένε καταχθάς ότι επανεκλέγεται ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Συγχαρητήρια κύριε Βαν Ρομπάι για τη συνέχιση της δραστηριότητάς σας. Πρέπει λοιπόν να σας συγχαρώ για αυτό. Αναφερθήκατε στο ότι οι αποφάσεις, αυτής, οι αποφάσεις αυτές ε, σηματοδοτούν αν θέλετε μία αλλαγή ε, μετά από αυτά τα οποία έγιναν. Δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ ε, θα έλεγα πιθανό σε λίγο καιρό η Ελλάδα να έχει ανάγκη πάλι από δισεκατομμύρια και για μια ακόμη φορά θα πρέπει να βρούμε αυτά τα δισεκατομμύρια και φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε καμία ουσιαστική προοπτική. Νομίζω λοιπόν ότι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συγκεκριμένη χώρας η Ελλάδα θα πρέπει να εγκαταλείψει τη ζώνη του ευρώ με διατεταγμένο τρόπο, με ελεγχόμενο τρόπο. Η Ελλάδα αυτή είναι φυλακισμένη σε μια νομισματική ένωση που δεν της επιτρέπει να είναι ανταγωνιστική μια επιπλέον προσπάθεια σωτηρίας δεν πρόκειται να βοηθήσει τίποτα. Αντί να κρατάμε ομήρους τους Έλληνες, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν λάθος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοζές δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε Βαν για τη νέα σας εντολή. Εγώ από την αρχή της θητείας σας Προσπαθώ να εξηγήσω στους συμπολίτες μου ότι η προσπάθειά σας είναι πολύ δύσκολη. Και το πιστεύω αυτό. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στους συμπολίτες μας. Λυπάμαι γιατί σήμερα πρέπει να πω ότι η Ευρώπη χάνει την αξιοπιστία της. Δεν αναφέρομαι σε εκλογικές μάχες εθνικού τύπου, εθνικής πολιτικής. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε γιατί τέτοιου είδους λόγια ε, γίνονται πιστευτά από την κοινή γνώμη. Γιατί η κοινή γνώμη ταυτίζεται με τέτοιες δηλώσεις εθνικού και εκλογικού τύπου. Γιατί φυσικά οι πολίτες μας δεν πιστεύουν στην Ευρώπη. Το πιστεύω στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αμφισβητείται. Χαίρομαι και θαυμάζω όλους αυτούς οι οποίοι Καθημερινά και κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα λένε τα ίδια πράγματα για την Ευρώπη, αλλά τα λόγια δεν φτάνουν. Οι πολίτες θέλουν λίγα λόγια και περισσότερες πράξεις. Θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Να δούμε τι φταίει σήμερα. Πρώτον, τα χρέη τα εθνικά τα οποία προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση και όλοι θα έλεγα δείχνουν μια εσωστρέφεια εθνική και δεν προσπαθούν συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λύσουν τα προβλήματα. Δεύτερον, η εξασθένηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ακούγεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δουλεύει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κανένας δεν ξέρει τι κάνει πραγματικά, γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί το πρόγραμμα δράσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες ε, να επιτρέψουν στον κόσμο να δει πώς πάνε τα πράγματα. Η Ελλάδα, η κατάσταση είναι δραματική. Γιατί πιστεύετε ότι ρυθμίστηκε το θέμα στην Ελλάδα. Όχι. Ρυθμίστηκε ένα επιμέρους πρόβλημα για να συνεχιστούν κάπως τα πράγματα. Αλλά σε ένα-δύο χρόνια τα προβλήματα ε, θα είναι πάντα μαζί μας. Και το διπλό πακέτο στο οποίο αναφερθήκατε προτείνω και μια ρήτρα σωτηρίας για τις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και μου είπατε όταν σας το είπα αυτό ότι όχι παρεμποδίζουμε την ελεύθερη λειτουργία των αγορών. Όχι. Πρέπει να μείνουμε στα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει και να εφαρμόσουμε αυτά που είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε. Κύριε Γκοζές, θέλει να σας θέσει μια ερώτηση ένα συνάδελφος. Yes, okay. Honorable one, prego. Ο κύριος Χουάνγκε θέλει να θέσει ερώτηση στον κύριο Γκοζές. Αγαπητέ συνάδελφε, αναφερθήκατε στη λαϊκή κυριαρχία ουσιαστικά και αναφερθήκατε επίσης και στο διπλό πακέτο για το οποίο μάλιστα είστε εισηγητής. Αναφέρομαι σε ένα ευρωπαϊκό θέμα. Λοιπόν, θέλετε να μεταφέρετε στην δευτερογενή ευρωπαϊκή νομοθεσία ένα κομμάτι της συνθήκης, αυτό, αυτή τη συνθήκη της λιτότητας, με αυτή τη ρήτρα η οποία θα μας βυθίσει, μια ρήτρα η οποία θα μας οδηγήσει στη μόνιμη ύφεση, όπως είπε και ο συνάδελφος Κονφά, πριν οι ίδιοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποφασίσουν για το αν θα επικυρώσουν αυτή τη συνθήκη. Εσείς που μιλάτε για λαϊκή κυριαρχία θα αποσύρετε την τροπολογία σας εννέα του, του, πακ, του διπλού πακέτου γιατί δείχνει να περιφρονεί τη δημοκρατία. Απαντά ο κύριος Γκοζές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στη συνθήκη ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνεί και ο κύριος Μπαρόζο λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει προτάσεις για να τα ενσωματώσει. Δεν αποσύρω τίποτα λοιπόν. Θεωρώ ότι η πειθαρχία η δημοσιονομική είναι απαραίτητη. Δεν χτίζει κανείς με φρούδες, ελπίδες και καλές ευχές. Πρέπει να συνδυάσουμε την ανάπτυξη και την πειθαρχία. Βέβαια την ανάπτυξη δεν θα τη βρούμε στη θεωρία και στα βιβλία, θα τη βρούμε στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εμπιστοσύνη. Αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Καλώς σας ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος Μάουρο. Συνάδελφος ε, Ενρίκε Γκουερέρο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια κύριε Φαν για την εντολή σας. Η, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συνομπουλίου εκτείνονται σε 12 σελίδες χωρίς μία γραμμή να αναφέρεται στις, στην ανίκεστο βλάβη που δημιουργείται από αυτές τις ε, πολιτικές και από αυτές τις ε, αποφάσεις. Η Ευρώπη είναι ένα μοναδικό μοντέλο ε, κοινωνικής αλληλεγγύης, έννοιας της ευρωπαϊκής ηθαγένειας πέραν των ε, οικονομικών χαρακτηριστικών της Ευρώπης. Το κοινωνικό μοντέλο πραγματικά υποφέρει όταν ασκείται επίθεση στα συνδικάτα, όταν υπονομεύεται ο δημόσιος διάλογος. Πράγματα που συμβαίνουν σε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία. Καταστρέφεται το τεράστιο πολιτικό εγχείρημα ε, της Ευρώπης από τους ηγέτες οι οποίοι προτιμούν να το καταστρέψουν τους ώστε να έχουν ελάχιστες ελπίδες να κερδίσουν τις ε, ε, εγχώριες ε, προεκλογικές τους μάχες. αντιμετωπίζουν την Ευρώπη οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τις τρομοκρατημένες εθνικές ε, απόψεις τους. Αυτό δεν είναι ε, πολιτική ηγεσία, είναι λαϊκισμός και καιροσκοπισμός και θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ. Ε, Ότι λόγω αν υποχρεώσεων ο κύριος Βαν Ρομπάι θα πρέπει να φύγει σε λίγο. Στις 10.50 θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μπαρόσο, στις 10.55 θα ακούσουμε τον κύριο Βον Ρομπάι. Προς το παρόν έχει το λόγο ο κύριος Όλε Σμίτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Α, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διατήρηση της Ενωμένης Ευρώπης μέσα από όλες αυτές τις εντάσεις είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για όλους μας. Ο πρόεδρος ε, Σαρκοζή θα έπρεπε να το σκεφτεί δύο φορές, πριν να πυροδοτήσει αυτές τις ε, εθνικιστικές συζητήσεις. Θέλουμε ε, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Αυτό είναι σαφές. Ωστόσο θα πρέπει να δίδουμε έμφαση στην ανάπτυξη, στην οικονομική μεγένθηση και χωρίως αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Το σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, να, να χτίσουμε μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων, να ε, οθήσουμε στην ανάπτυξη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό βεβαίως πρέπει να αρθούν τα ε, φορολογικά εμπόδια. Θα αφήσουμε μια γενιά ολόκληρη, μια ολόκληρη γενιά χωρίς καμία προοπτική. Και ήθελα να πω το εξής και μάλιστα στα αγγλικά προς τον κύριο Γκόλνης και τους λοιπούς. Καλό θα ήταν να υπενθυμίζουμε συχνά περί τίνος πρόκειται ε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ε, ποια είναι η ευρωπαϊκή ιστορία μας. Ε, η ιστορία διδάσκει κύριε Γκέλνης ότι στο παρελθόν λύναμε τα προβλήματά μας στα πεδία των μαχών. Πλέον δεν το κάνουμε πια. Εγώ ακούω εσάς και εσείς ακούτε εμένα. Αυτό τον τρόπο θα πρέπει να προτιμούμε ε, πλέον. Νομίζω ότι στίγεται ε, αυτή την ευρωπαϊκή ιδέα συνεργασίας, την καταστρέφεται, καταφέρετε βαρύ πλήγμα εναντίον της και θα πρέπει να αναλάβετε τις δικές σας ευθύνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Σουίνμπερν, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Στο μέλλον θα είναι σωστό όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο αρχικό σύμφωνο σταθερότητα να υιοθετηθούν από όλε τι κυβερνήσει. Όταν όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, αναγνωρίζουμε ότι οι κυρώσει και τα πρόστιμα λειτουργούν μονάχα όταν έχουν επανέλθει σε επίπεδο σταθερότητα οι χώρε και ιδίως σε οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι πολύ αφελές από τον Κομισιόν να μην συμφωνεί με την Ισπανική κυβέρνηση για τις διαστορικές αλλαγές και τη μείωση του ελλείμματος. Η δήλωση του Ισπανικής κυβέρνησης για το 2% του κρατικού ελλείμματος θα ε, καταστήσει τους στόχους αρχικούς αδύνατο να επιτευχθούν εάν παρέμβει η Κομισιόν όπως το κάνει. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη που θέλουν πραγματικά μεταρρύθμιση να έχουν χρόνο και δυνατότητες να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους των, για αυτές ιδανικότερο τρόπο. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να πάρει τα ειδικά μέτρα για να επανέλθει σε οικονομική υγεία. Δεν θα πρέπει να υποσκάψουμε την αξιοπιστία των νέων κοινοτικών κανόνων. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Γιώργιν Κλούτε έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παρόζο, κύριε Φανουλαπόη, ποια είναι η μορφή που έχει για τους πολίτες η επεξεργασία της κρίσης μετά την τελευταία διάσκεψη κορυφής. Βλέπουν ότι παίρνουν οι τράπεζες ένα δις από την ε, κεντρική τράπεζα χωρίς όρους και μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά όπως θέλουν. Οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση όμως καταδικάζονται σε μια καταστροφική πολιτική λιτότητα. Είναι αναγκασμένη να εγκαταλείψουν τους μισθούς τους, τις ε, συντάξεις τους ε, και να υπάρχουν περικοπές στα κοινωνικά θέματα. Εν αντιθέσει όμω προ τη Γερμανία, οι οικονομίε των χωρών αυτών δεν εξαρτώνται από τι εξαγωγέ, αλλά από την εσωτερική αγορά των εν χωρών. Και αυτέ οι εσωτερικέ αγορέ καταστρέφονται από την υποχρεωτική αυτή πολιτική λιτότητα. Κύριε Μπαρόζο και Ρουμ Φαρόμπα, δεν βγαίνει κανένα έτσι να μπορεί το να βγει από την κρίση, απλώ θα έχει πληρή αποτυχία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριο Συνοκόρας Αλαβράκο κύριε πρόεδρε φοβάμαι ότι με αρκετή αοριστία μιλάμε για ανάπτυξη ενώ δίνουμε κύρια σημασία στη δημοσιονομική πειθαρχία που όμως από μόνη της δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να επιλύσει. δεν πρέπει να ξεχνάμε οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. παράλληλα αναγνωρίστηκε ότι η φοροδιαφυγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο διωγγούται και δεν ελέγχεται ενώ το ασφαλιστικό σύστημα είναι η επόμενη βόμβα που θα συνθλίψει το σύστημα. η ανεργία τίνει να πάρει μορφή χιονοστιβάδας. το μήνα δεκέμβριο το ποσοστό ανεργίας στην ελλάδα έφτασε το 21% και ένας στους δύο νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών είναι άνεργος. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κορμό της κοινωνίας κλείνουν η μία μετά την άλλη. τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζονται σε όλες σχεδόν τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και ο κοινωνικός εστός της ευρώπης απειλείται. κύριε βαν ρομπάι σας συγχαίρω για την ανανέωση της εντολής σας και θέλω να πω σε εσά και στον κύριο μπαρόζο ότι δεν πρέπει να περιμένετε να σας συγχαίρουν διότι το συγχαίριν είναι χαλεπότερο το συλληπίστε. κάντε τη δουλειά σας και προχωρήστε μπροστά. ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Βέρτμαν έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις ε, περασμένες ε, ε, διασκέψεις κορυφής έγιναν σημαντικά βήματα για να προχωρήσει η Ευρώπη προς μια άγουσα ανάπτυξης ε, και σταθερότητας. Παραδείγματος χάρη ε, το διτό αυτό, τα δύο αυτά μέτρα, το Stuttgart θα πρέπει μας για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους του 2020 θα πρέπει να προχωρήσουμε, να προωθηθεί η εσωτερική αγορά και να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Έχω σημαντικέ όμω ε, επιφυλάξεις όσον αφορά την ανεργία των νέων. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα, του δώσει να μειώσουμε τα σημα... σημερινά στοιχεία και να δώσουμε καινούριε ευκαιρίε στους νέου. Μου φαίνεται ότι οι επενδύσει στην παιδεία και μετεκπαίδευση είναι η καλύτερη προπόθεση για να υπάρχουν Νέε ευκαιρίε. Α δώσουμε στους νέου μα αυτή την ευκαιρία. Δικαίωμά τη είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σάιβελ Βόλσκι, δύο λεπτά. Νομίζω ότι ο καιρό περνάει. Περνάει μάλιστα μεγαλύτερη ταχύτητα από τις συναντήσεις του Συμβουλίου. Για την οικονομική κρίση ακούστηκαν τα πάντα αλλά οι δράσεις για να αντιμετωπιστεί δυστυχώς είναι ανεπαρκής. Χρειαζόμαστε φυσικά και σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να πάρει αποφάσεις για κυρώσεις, για πειθαρχία, αλλά δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις για την ε, ανάπτυξη. Μου θυμίζει λίγο τις αποφάσεις για την οικονομική ανάπτυξη ε, στις σοσιαλιστικές χώρες θα πρέπει να υπάρξουν αναπτυξιακά ομόλογα χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξεχνάμε το πλαίσιο της κρίσης. Μια συλλογική κόποση αν θέλετε ε, από τη μία των ευρωπαϊκών χωρών και μια ανάπτυξη των εθνικιστικών θα έλεγα αισθημάτων. Και αυτό φαίνεται και στα πλαίσια του διαδικτύου Νομίζω ότι τέτοιου είδους ε, ιδέες παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, είναι οι πλευρικές θα έλεγα ζημίες, επιπτώσεις στις, ε, στην υπόλοιπη οικονομία του κόσμου η οποία δεν ενισχύεται από την κατάστασή μας και επίσης και στο Σέγγεν το οποίο και αυτό κλονίζεται. Για την Ελλάδα τώρα. Έγινε μια θαυμαστή προσπάθεια διάσωσης της όχι μόνο για την ίδια την Ελλάδα, αλλά στα πλαίσια της αλληλεγγύης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολιτική σημασία έχει η προσπάθεια αυτή. Η Ελλάδα δεν τα πάει καθόλου καλά οικονομικά. Είναι η χειρότερη οικονομία από όλες τις χώρες. Τα ίδια θα μπορούσε να πει κανείς όμως και για την Ουγγαρία, η οποία τιμωρείται ουσιαστικά για την ε, καταστροφική οικονομική κατάσταση την οποία άφησε, στην οποία άφησε τη χώρα η προηγούμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση και την τιμωρείται διπλά. Σήμερα η Ισπανία ας πούμε μπορεί να μην εφαρμόσει τους στόχους μας αλλά η Ουγγαρία τιμωρείται ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για τα ελλείμματα. Τι μηνύματα θέλετε να στείλετε εσείς σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν το καλό και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να το κάνουν. Η πολιτική σας δεν είναι συνεκτική, δεν είναι η σωστή. Ευχαριστώ συνάδελφε, η κυρία Περβάνς Περές. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Να μεταφέρω ένα μήνυμα στον πρόεδρό μας. Να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ για την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ήταν σημαντική η παρουσίασή του. Έθεσε σε αντίθεση την ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πρότυπο και από την άλλη για το πόσο δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Το Συμβούλιο αυτό χαρακτηρίστηκε από την υπογραφή μιας συνθήκης. Αν και μία από τις κυβερνήσεις που είναι υπέρ της στρατηγικής Μερκοζή, στην ουσία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Ούτε η Ισπανία ούτε οι κάτω χώρες δεν θα εφαρμόσουν αυτά τα οποία υπέγραψαν. Αν κατάλαβα επίσης πρόεδρε, ξαφνικά οι υπευθύνοι ανακάλυψαν ότι πρέπει να μιλήσουμε και για την ανάπτυξη. Ε, βέβαια όχι με τον ίδιο τρόπο. Όχι με χρυσούς κανόνες, αλλά με κανόνες ολίγων, θα έλεγα, θολούς. Και όμως ανάπτυξη δεν θα υπάρξει αν δεν εφαρμόσουμε παρά μόνο τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, που είναι κανόνες που θα τους κατήριζα κανόνες εσωτερικής αρνητικής ανάπτυξης. Εσείς στην ουσία συστηματικά αλλάζετε απόψεις. Δεν θα οδηγήσετε στην ανάπτυξη με την καταστροφή του ευρωπαϊκού προτύπου. Υπονομεύετε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πρέπει να σκεφτείτε πρώτα απασχόληση, κοινή βιομηχανική στρατηγική, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στα θέματα της ενέργειας, κοινοί τρόποι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καταγγελία των μονομερών πολιτικών των κρατών μελών. Εάν δεν υπάρξει συνοχή ανάμεσα στα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των πολιτικών που έχουν προαποφασιστεί επί τη βάση των ιδίων πόρων, επί τη βάση των νέων ομολόγων και επί τη βάση μιας σωστής φορολογικής πολιτικής. Θα μεταφέρω αυτό που είπατε στον πρόεδρο Σούλτς. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπαρόσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Απαντώ συγκεκριμένα στα ερωτήματα που ετέθησαν. Καταρχήν, όσον αφορά την επιστολή των 12 ε, κυβερνήσεων. Είπα στη διάσκεψη κορυφή ότι θα μπορούσα να συμφωνήσω σχεδόν με κάθε λέξη τη επιστολή αυτή. Ήταν όλα στοιχεία πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη. Ενδυνάμωση της εσωτερική αγορά, και διορθωτικές μεταρρυθμίσει. Υπενθύμιζε όμως επίση τα κράτη-μέλη δύο πτυχέ που μου φάνηκαν σημαντικέ. Πρώτον, ότι στην επιστολή αυτή δεν γινόταν καμία αναφορά στην ε, κοινωνική διάσκεψη, ε, διάσταση και την ανάγκη καταπολέμηση της φτώχειας. Θα πρέπει διαρθρωτικά μέτρα να συνδεθούν με ενεργά μέτρα ε, για την κοινωνική διάθεση. Επίσης τόνισα την έκπληξή μου ότι δεν υπήρχε μία, μία μόνη αναφορά στη στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Δηλαδή, μία στρατηγική που ενεκρίθη ομοφωνά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αναφέρεται καν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και γι' αυτό κάνω και εδώ μια έκκληση στο Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε μια στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμόσουμε. με αποφασιστικότητα όλες τις πτυχές. Αυτό είπα όταν αναφέρω ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα. Στην απάντηση που έστειλα στους 12 αρχικούς και κυβερν... Ε, κρατών και κυβερνήσεων ε, ένα παράρτημα που αναφέρεται σε όλες τι προσπάθειε που κατεβλήθησαν από τα θεσμικά όργανα, όχι δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόνο, αλλά και από το Κομισιόν και το Συμβούλιο και βλέπουμε ότι ορισμένα από τα θέματα έχουν μπλοκάρει ακριβώς από κυβερνήσει που υπέγραψαν. Παραδείγματο χάρη. Το δίπλωμα ευρεσυλλεκτία, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσυλλεκτία συζητιέται εδώ και 30 χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τώρα κυβερνήσει που καλούν την Ευρώπη να κάνει περισσότερη για την ανάπτυξη, εξακολουθούν όμω να παρεμποδίζουν αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσυλλεκτία. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε όταν λέμε Ευρώπη. Όταν λέμε η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή δυσκολίες. Λυθέ. Θα πρέπει να δούμε ποιο καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προωθηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο και ποιο πολλές φορές μπλοκάρει τις εξελίξει, Αυτό είναι ένας όρο εκ των ανεφ για να υπάρχει μια δίκαια πολιτικά αλλά και πνευματικά συζήτηση. Όσον αφορά την Ελλάδα. Ακριβώς εδώ χρειάζεται τιμιώτης. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση λόγω του ευρώ. Γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες εκτός ευρώ που χρειάζονται επίσης προγράμματα ενίσχυσης. Και χώρες μάλιστα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σκέφτομαι εδώ την Ισλανδία που έχει επίσης τεράστια προβλήματα παρόμοια με μια γενική κρίση πληρωμών. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι κυρίως το αποτέλεσμα δύο αιτιών. Καταρχήν, η συνεχής αύξηση του δημοσίου χρέους σε πολλούς χώρους και επίσης η ανευθυνότητα της ε, συμπεριφοράς σε πολλούς τομείς ε, δημοσιονομικούς και εντός και εκτός ε, ενώσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ προβλήματα που είναι δύσκολο να επιληθούν γιατί είμαστε μια νομισματική ένωση που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τα μέσα της ε, Οικονομικής Ένωσης και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά είναι εσφαλμένο, πλήρως εσφαλμένο να πούμε ότι η σημερινή κρίση είναι η επίπτωση του ευρώ. Ε, των αντίον, ίσως το ευρώ είναι η λύση της σημερινής κρίσης. Γι' αυτό εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να δεχτώ ορισμένους που έρχονται εδώ και λένε ότι λυπούνται τόσο για όσα υποφέρει η Ελλάδα, ότι λυπούνται για όλες τις δυσκολίες που έχει η Ελλάδα, αλλά η δική τους κυβέρνηση δεν ξόδεψε ούτε ένα ε, λεπτό, ούτε ένα ευρώ για να βοηθήσει την Ελλάδα. Και τι προτείνετε σαν λύση για την Ελλάδα, πτώχευση, πτώχευση, πτώχευση για να μου εξηγήσουν γιατί η χρεοκόπηση ενός, χώρου, ε, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η λύση. Πώς θα υπάρχει η εμπιστοσύνη στις χώρες αυτές για επενδύσεις. Πώς η παράλυση του, του δημοσίου τομέα της χώρας αυτής, ε, η ε, κατάρρευση των σχολείων, των νοσοκομείων θα είναι η λύση για τη χώρα αυτή. Σας παρακαλώ, ας είμαστε σοβαροί είναι πραγματικά άτιμο πολιτικά και πνευματικά να λένε ότι η πτώχευση είναι η λύση για τα προβλήματα της Ελλάδας. Άλλοι λένε ότι τα προγράμματα αυτά δεν θα λειτουργήσουν. Ότι είναι έμπνευση της Τρόικα. Για να είμαστε όμως σοβαροί. Το πρόγραμμα για την Ελλάδα είναι το πρόγραμμα που εγκρίθηκε ομοφωνά από τα κράτη-μέλη της ζώνης ε, ευρώ και όλοι έδρασαν μέσα στα πλαίσια της εντολής που είχαν από εκεί και πέρα. Λοιπόν, όλοι εκείνοι που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα που ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα το ενέκρινε όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η Βουλή με τα δύο κύρια κόμματα. Αντί λοιπόν να λένε να δεν θα λειτουργήσει, ας μας βοηθήσουν να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει τεράστιο κόστο. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα του βοηθήσουμε να επομιστούν κάποιο κοινωνικό ε, άκτο που θα είναι τεράστιο. Αλλά το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να προωθηθούν οι διαστατικέ μεταρρυθμίσει για να μπορέσει η Ελλάδα να κερδίσει την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται. Ένα άλλο θέμα που ετέθηκε για τα πρότυπα που ξαναναφέρθηκε από το φίλο Σάριου Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση. Η Κομισιό θα επιβάλλει τις συνθήκες ή ε, ισότιμα και χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτά που είπατε για την ε, ε, Ισπανία και τη Γαλλία δεν είναι σωστά ή και σε σχέση με την Ουγγαρία γιατί θα έπρεπε η Ουγγαρία να έχει φτάσει στη μείωση του ελλείμματος το 2011. Η Ισπανία το 2013. Προτείναμε στην Ουγγαρία κάποια μέτρα. Αλλά όχι μόνο στην Ουγγαρία. Πέντε χώρες είναι εκείνες στι οποίε υποβάλαμε τι προτάσεις. Η Πολωνία, η Κύπρος, η Μάλτα, το, Βέλτιο, το Βέλγιο και η Ουγγαρία. Όλοι δέχτηκαν τα μέτρα αυτά εκτό από την Ουγγαρία. Δεν έτυχε λοιπόν η ειδική μεταχείριση στην Ουγγαρία η Ουγγαρία δεν θέλησε να ακολουθήσει και να δεχθεί τις προτάσεις που έκανε η Κομισιόν. Εν αντιθέσει με αυτό που έκανε η Πολωνία, η Κύπρος, η Μάλτα και το Βέλγιο. Και σας το λέω αυτό ειλικρινά γιατί θα ήταν ένα σφάλμα να υπάρχει τώρα ένα χάσμα μεταξύ των χώρων που βρίσκεται εντό και εκείνο που είναι εκτός της ε, ζώνης ευρώ. Η Κομισιόν πάντα προάσπισε την ενότητα της Ευρώπης. Δεν θα έχουμε τώρα δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάλογα που βρίσκεται κάθε χώρα. Τελικά όμως, μέσω των πολύ χρησίμων στοιχείων της συζήτηση είδα ότι υπάρχουν κάποια σημεία συναντικά, τουλάχιστον μέσα στις πιο ισχυρέ ε, πολιτικές δυνάμεις. Καταρχήν, ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων μέσα στα πλαίσια των ομάδων δράσης που δημοσίσαμε θέλει, πρέπει να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Και θέλω να πω εδώ στους βουλευτές ότι η Κομισιόν δεν κάνει μόνο δηλώσεις, έκανε ήδη συγκεκριμένε προτάσεις. Υπάρχει η πρωτοβουλία μας για την οδηγία για τις ε, αποταμιεύσεις και θα πρέπει επίσης να σας πω ότι ζητήσαμε μια, με μια πρόταση μια εντολή διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες που βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου εδώ και μήνες και μπλοκάρεται από δύο χώρες. Και ξέρετε ότι χρειάζεται ομοφωνία. Λοιπόν, μην κατηγορείτε την Κομισιόν να κατηγορήσετε αυτές τις δύο χώρες που μπλοκάρουν. Και για την Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι αυτό ήταν ένα από τα θέματα της συζήτησης μου με τον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήμου και με άλλα μέλη της Κομισιόν. Τους κάλεσα δηλαδή ακόμα και πριν να υπάρχει ε, μια συμφωνία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για, με την Ελβετία και με άλλους θα πρέπει η Ελλάδα να έχει μια διμερή συμφωνία με την Ελβετία. Όχι μόνο το ανέφερα αυτό στον Έλληνα Πρωθυπουργό, το είχα ήδη αναφέρει στην πρόεδρο της ε, Ελβετίας την περασμένη φορά που την είδα. Κάτι άλλο που είδα να ε, υπάρχει εδώ συνένεση είναι η ανάγκη ε, ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Και ήδη ανακοίνωσα ότι το φθινόπωρο θα υποβάλει η Κομισιόν το νόμο της ενιαίας αγοράς. Μπορείτε να βαστείτε ότι θα το κάνουμε. Ο τρόπος για να συμπληρώσουμε τις δράσεις μας με επενδύσεις και γι' αυτό υποβάλαμε στην Τράπεζα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάποια πρόταση για τα ομόλογα ανασχέδιο, όπως λέγονται, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Υπάρχει συμφωνία πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν οι πόροι για αυτές τις επενδύσεις. Οι περισσότερες χώρες μελή δεν έχουν περιθώρια ελιγμών για αυτού του τύπου τη επενδύσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν και συμφωνούν εδώ οι μεγάλε πολιτικέ ομάδε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε να βρούμε κάποιου πόλου για τι επενδύσει αυτέ ή με τα project bonds αυτά ή με τι μελλοντικέ χρηματοπιστωτικέ προβλέψει και ελπίζω ότι θα συνεργαστεί η την Κομισιόν να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα βάσει των φιλοδοξιών μας γιατί πραγματικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι μοχλοί ανάπτυξης ε, καινοτομία, έρευνα και άλλα ευρωπαϊκά μέσα. Όλα αυτά θα επιτύσσουν πολλή εργασία, πολλή αποφυστικότητα και πραγματικά πιστεύω ότι για ανάπτυξη της Ευρώπη δεν χρειαζόμαστε περισσότερες εξαγγελίες δεν θα πετύχουμε έτσι ανάπτυξη, αλλά μόνο αν είμαστε σοβαροί κατά την εφαρμογή εγγυούμενοι κάθε φορά ότι είμαστε θέση να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις και τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του ε, Κομισιόν, πρόεδρος του Συμβουλίου. Κύριος Φανερόπα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω ε, για τα συγχαρητήρια που εκφράσατε για την επανεκλογή μου ε, στο ε, αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διαπίστωσα ότι δεν είναι όλοι το ίδιο ενθουσιώδης. Ωστόσο αυτό είναι θεμητό ασκήθηκαν επικρίσεις για τη στρατηγική μας, για τη γενικότερη προσέγγισή μας. Θα ήθελα να το, σχολιάσω αυτό, να το σχολιάσω αυτό. Η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει και σε επίπεδο ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι μια στρατηγική που έτυχε τη στήριξη των πάντων, όλων των κρατών μελών, όλων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από το ξέσπασμα της κρίσης από την αρχή της πριν από δυόμιση χρόνια. Και μάλιστα και σε διαφορετική σύνθεση, γιατί ξέρετε αυτοί που με εξέλεξαν πριν από δυόμιση χρόνια ε, πολλοί έχουν φύγει και έχουν μείνει πλέον 12 από, τους, ε, ε, από το σύνολο όλα και τα 27 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Μπορεί κανείς να επικρίνει αυτή τη γενική προσέγγιση, το μόνο που απαντώ εγώ είναι ότι αυτή είναι μια συνολική ομόφωνη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ε, πολύ δύσκολος αυτός ο δρόμος. Δεν την χάνει λαϊκή στήριξη. Παράγει αποτελέσματα μόνο μέσω πρόθεσμα, αν όχι και μόνο μακροπρόθεσμα ε, τελικά. Όμως αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε διαλέξει και θα ε, επιμείνουμε στην επιλογή μας αυτή. Κατά τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις είπα ότι η στρατηγική μας θα λειτουργήσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Νομίζω ότι πάντοτε οι δηλώσεις μου είναι πολύ μετριασμένες. Εγώ πάντοτε μιλώ με πολύ μετριασμένο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι είναι το τέλος της κρίσης. Μίλησα για σημείο καμπής και νομίζω ότι παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις μου. Είναι θετικό το γεγονός ότι στον τύπο δεν γίνεται πια λόγος για το τέλος της Ευρωζώνης. Αυτό ακριβώς εννοώ. Βεβαίως και δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Ωστόσο, όταν βλέπω ότι η διατραπεζική αγορά αναζωπυρώνεται, όντας νεκρή εδώ και μήνες, όταν βλέπω διάφορα θετικά στοιχεία σε διάφορα επίπεδα, τότε ε, δικαιούμαι πιστεύω να πω ότι πράγματι έχουμε καλύψει, έχουμε φτάσει στην κορυφή της ανηφόρας και παραμένει ε, ένας επίπεδος δρόμος που θα πρέπει να διανύσουμε πριν πάμε πλέον σε πιο κατηφορικό και εύκολο έδαφος. Από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ευρωζώνης. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πρώτη και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο μέλλον της Ευρωπο... Ε, Ευρωζώνης. Αυτό είναι το βασικό και θα είναι το πρόδρομο σημάδι για την επιστροφή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το, η ένδειξη δηλαδή πλέον ξανά εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη είναι σημαντικές. Γίνεται λόγος για τα firewall, γίνεται λόγος για τις διάφορες πρωτοβουλίες ε, περί της δημοσιονομικής σταθερότητας και των οικονομικών του κράτους. Πέρα από όλα αυτά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το πιο σημαντικό είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά της απασχόλησης και στην αγορά των προϊόντων και δεν το έχουμε συζητήσει επαρκώς εδώ. Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Αυτά χρειαζόμαστε, αλλιω η κρίση θα μας ξαναπλήξει αργά ή γρήγορα. Αυτό το οποίο με εξέπληξε εδώ ε, σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι κανείς δεν αναφέρθηκε ούτε ε, για μία φορά ε, στους όρους ευαικό εξάμεινο. Ενδεχομένως κάποιοι το υπενήχθηκαν τρόποτινά, αλλά κανείς δεν το ονομάτισε καν από εσάς. Αυτός ήταν ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να αξιολογήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, να δει ε, πού ακριβώς βρισκόμαστε και σε επίπεδο τήρησης των προϋπολογισμών και σε μακροοικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ε, θέσεων απασχόλησης και πολιτικών απασχόλησης. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα σχέδια σταθερότητας για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και τον Μάιο και στη συνέχεια στο Συμβούλιο του Ιουνίου θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά την έννοια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τότε αργά ή γρήγορα η κρίση θα ξεσπάσει και ξανά. Εκφράζω την απογοήτευσή μου, διότι κανείς δεν σχολίασε αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα το οποίο έχουμε εγκρίνει τόσο ενθουσιοδός εμείς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μεγάλη πρόκληση για όλους μας είναι η εξή. Σε περίοδο αναπόφευκτης εξυγίανσης των δημοσιονομικών σε σχεδόν όλων, όλες τις χώρες οφείλουμε ε, να διατηρήσουμε τις μακροπρόθεσμες ε, πολιτικές μας προκειμένου να πετύχουμε τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 πέρα και ταυτοχρόνως με την εξυγίανση των δημοσιονομικών, προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι βεβαίως να εξαλείψουμε τα ελλείμματα και να μειώσουμε το χρέος, διατηρώντας ωστόσο τις ελπίδες για το μέλλον και διατηρώντας τις δαπάνες και τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης των νέων, διατηρώντας τις επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν εν μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανση να διατηρηθούν και αυτές οι επενδυτικές προτεραιότητες. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση, πώ θα καταφέρουμε να συγκεράσουμε τα δύο. Εξού και ε, ζητήσαμε τη γιγάντια συνεισφορά των τραπεζών. Ε, χάνουν το, αυτή τη στιγμή ε, το 70% της ονομαστικής αξίας του ελληνικού χρέου, χρέους προκειμένου να εξυγιανθούν τα οικονομικά της χώρας αυτής. Συμφωνώ με όσους ζήτησαν την υιοθέτηση ακόμα πιο αυστηρών μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Έχουμε τον κανόνα της ομοφωνίας ε, για το φορολογικό καθεστώς. Η Επιτροπή έχει πολλές προτάσεις να υποβάλει. Πολλά μπορούν να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Ξέρετε, ε, ε, εάν ένα πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα είναι η αδυναμία ίσπραξης ε, βεβαιωθέντων φόρων. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η τεράστια κοινωνική αδικία και είναι και η πηγή του τεράστιου δημοσίου ελλείμματος το οποίο εμφανίζει η χώρα αυτή. Οι πολιτικές εξοικίανσεις των δημοσιονομικών θα πρέπει να συνοδεύονται από δράσει στήριξη τη αλληλεγγύη. Και γι' αυτό το λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς αποφασίσαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και η βοήθεια που της προσφέραμε ανέρχεται στο 100% του εθνικού ε, του εγχώριου, ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας αυτής. Είναι ε, νομίζω πολύ εύγλωτοι η αριθμοί. και θα πρέπει εν μέσω πολιτικής εξοικείανσης των δημοσιονομικών θα πρέπει ε, να μην ε, χάνουμε από τα μάτια μας τους στόχους τους κλιματολογικούς ε, τους στόχους επίτευξης ενεργειακής αποδοτικότητας. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη για άλλη μια φορά, ε, πέρα από τη δημοσιονομική εξυγίανση, να υιοθετήσουν συγκεκριμένε πολιτικέ για την απασχόληση. Εξού και με μεγάλη ανεπομονησία ε, περιμένουμε το σχέδιο για την απασχόληση ε, σε κάθε κράτο μέλο, το οποίο θα υποβληθεί στο αντίστοιχο Συμβούλιο του Απριλίου και θα στηριχθεί στις συστάσεις της Επιτροπής και θα συζητηθεί ξανά τον Ιούνιο. Τώρα, είναι σαφές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργό έχει αναλάβει ε, πολύ μεγάλες δεσμεύσεις ε, για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στην Ελλάδα. Η εμβάθυνση στην, της αγορά, αγοράς, της εσωτερικής αγοράς είναι κάτι που μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω κονδύλια. Έχοντας διαβάσει προσεκτικά ε, το περιεχόμενο των τελευταίων σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, σχεδίων ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να πω ότι δεν χρειάστηκε καν να το συζητήσουμε. Ε, με την επιστολή των 12 ε, είχαμε ένα αποτέλεσμα ευρεία συνένεσης και συμφωνίας. Τώρα, ως προς την αναζωπήρωση των οικονομιών μας, έχω να πω το εξής η περίοδος κατά την οποία πυροδοτούσαμε την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω ε, της δημιουργίας υπερβολικών χρεών έχει πλέον παρέλθει. Χρειάζεται μια πιο ε, εκλεπτισμένη προσέγγιση, μια πιο προσεκτική προσέγγιση διατηρώντας σε χαμηλό επίπεδο τις δαπάνες αλλά ε, και διατηρώντας ωστόσο ε, σε ικανοποιητικό επίπεδο τις δαπάνες που μπορούν να οδηγήσουν στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Τώρα, ως προς την Συρία και τη Βοσνία. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουμε την εντολή από πλευράς ε, Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι οι χώρες ε, οι ευρωπαϊκές που μπλοκάρουν την κατάσταση. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Εξετάσαμε τις διάφορες επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας ως προς το θέμα της Συρίας. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Θέλουμε να ε, υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά για να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουμε μας χρειάζεται εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη λάβαμε αυτή την ε, εντολή για τη Λιβύη, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά δεν την έχουμε λάβει ακόμα για τη Συρία προκειμένου να αυξήσουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια εκεί. Ως προς τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ε, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον νέο ε, Πρωθυπουργό και εξετάσαμε τις, τους προσανατολισμούς, τους φιλοευρωπαϊκούς προσανατολισμούς της ε, ε κυβέρνησης αυτής. Είδαμε ότι θεωρούν ότι το μέλλον τους βρίσκεται στην Ευρώπη και θέλουμε ε, να προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική στη χώρα αυτή. Πρώτη φορά ε, βλέπουμε ε, να εκφράζεται φιλοευρωπαϊκή πολιτική βούληση στη χώρα αυτή η οποία πράγματι έπαιξε ένα τόσο τραγικό ρόλο στον πόλεμο που ξέσπασε στην επικράτειά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φενροπόη. Είπατε ότι ενθουσιασμός για την επανεκλογή σας εκφράστηκε σε, με διαφορετικό τρόπο εδώ είναι νομίζω φυσιολογικό αυτό. Ε. Ένα ετερογενές ε, κοινοβούλιο εκφράζει διαφορετικά τον ε, ενθουσιασμό του, αλλά το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σα συγχαίρει για την επανεκλογή σα. Να είστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο σα και θα ήθελα από εδώ να πω ότι η δική σα προσωπική στάση και η εντύπωση που μας δίνεται σε όλο το σώμα μας έχει εντυπωσιάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω τώρα μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τους ε, πρόεδρους κυρίους ε, Φανταπάη και Μπερόζο. Καλύτερα να έμεναν εδώ, αλλά δεν θέλουν. Ας ε, δουν τι θα καταλάβουν. Ο συνάδελφος Χάκλοντ έχει το λόγο. Κύριε Βαν Ρομπά, κύριε Μπαρόσο που φεύγετε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι οι θέσεις απασχόλησης δεν μπορούν να βασίζονται στα ελλείμματα και στα υπερβολικά εθνικά δημόσια χρέη. Χαίρομαι που το άκουσα αυτό για μια ακόμη φορά και χαίρομαι γιατί ο κύριος Βαν Ρομπάι αναφέρθηκε στο λεγόμενο εξαπλό πακέτο έχουν γίνει πολλά χάρη σε αυτό το πακέτο. Είναι λυπηρό που η Ουγγαρία δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το διπλό πακέτο, το 2-pack, καλό θα ήταν και το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι απαιτείται μεγαλύτερος αυτοματισμός για να έχουμε αποτελεσματικότητα. Ήταν εναντίον το Συμβούλιο σε αυτό τον αυτόματο χαρακτήρα ο κύριος Φερχώστα τα αναφέρθηκε και στο Ταμείο Σωτηρίας. Αν δεν το κάνουμε αυτό τότε φοβάμαι ότι θα ενισχύουμε τους μηχανισμούς σωτηρίας χωρίς όμως να καλύπτουμε τις ανάγκες των αγορών. Για την στρατηγική 2020 και αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπαρόσο να θυμίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου το ίδιο το Συμβούλιο ήθελε να κόψει 560 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα από τον επόμενο προϋπολογισμό. Το, το Κοινοβούλιο ευτυχώς το γλίτωσε σε εισαγωγικά, γλίτωσε αυτή την περικοπή, αλλά αυτό δείχνει το πνεύμα ορισμένο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ επόμενος για δύο λεπτά, Presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι η τρίτη φορά που παίρνω το λόγο στην Ολομέλεια ως προς το θέμα αυτό. Και λυπούμε διότι θα επαναλάβω αυτά που έχω πει ε, ξανά. Όπως έλεγε ο Μικέλντε Ουναμούνο, ε, που είναι ένας μεγάλος Ισπανός συγγραφέας, ο μόνος τρόπος να ε, πριονίσει κανεί ένα δέντρο όταν πρέπει να το κόψει είναι σιγά σιγά σιγά σιγά να ε, πριονίζει τον κορμό. Με μικρά χτυπήματα δηλαδή ε, καταφέρνετε το μεγάλο πλήγμα που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε απασχόληση, χρειαζόμαστε δουλειά κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Ε, με τη λιτότητα μπορεί να έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά δεν, ξε, αλλά θα πρέπει να φύγουμε από την κρίση για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ευημερία. Επιγόντως θα πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα για την αναζωπήρωση της ανάπτυξης και όλα αυτά τα μέτρα έχουν συμφωνηθεί στα τελευταία Ευρωπαϊκό Συμβούλια και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις. Η Ισπανία έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση ε, για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Σε λιγότερο από 100 μέρες έχουμε υιοθετήσει τρεις μεταρρυθμίσεις κλειδιά. Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Και θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Όπως λέει και ο Μαριάνο Ραχόη, η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν αναγγέλει μόνο μεταρρυθμίσεις, αλλά τις υλοποιεί κιόλας, κάτι το οποίο δεν είναι το ίδιο με την αναγγελία βεβαίως η υλοποίηση. Κάθε φορά που ανακοινώνουμε σχέδιο θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε. Ε, για να... Ε, ε, προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις. Όπως είπε και προσφάτως ο, ο πρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης, ο Μαριάνο Ραχώη και όπως ε, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Λουίς Ντεκίντος, η Ισπανία εκπληρώνει τις ε, υποχρεώσεις της και θα τις εκπληρώσει και στο μέλλον. Έχουμε υιοθετήσει μια στεναρή στάση υπέρ της Ευρώπης. Δείχνουμε τα χαρτιά μας, είμαστε ειλικρινείς και ε, πρόκειται να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις στο ακέραιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Είδατε ότι έχουμε μια καθυστέρηση χρόνου και γι' αυτό θα πρέπει να είμαι δυστυχώς πολύ αυστηρός στο τα χρονοβόρευσης. Πιο αυστηρός ότι η προκατοχή μου. Εν τω μεταξύ έχουν αναβληθεί νομίζω οι ψηφοφορίε για τις μία. Στόλφος Μπούλμαν έχει το λόγο, δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, προγράμματος στην πραγματικότητα της οικονομικής εξέλιξης. Αρχές ε, του χρόνου ε, μειώθηκε το, η ανάπτυξη στην, Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία το ίδιο, στην Πορτογαλία η εικόνα δεν είναι πολύ καλή, στις κάτω χώρες υπάρχει ε, το πρόβλημα και ακόμη και στη Γερμανία μειώνονται οι, ο τζίρος των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκαν 10 15 φορές στους όρους ανάπτυξη και ε, απασχόληση. Και τι άλλαξε από το είπανε, τίποτα. Το να λένε και να ξαναλένε τα ίδια δεν αλλάζει τίποτα. Θέλω λοιπόν να ξέρω τι είναι το καινούριο τώρα και στην ενασχόληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Κομισιόν. Ο κ. Μπαρόζο ανέφερε κάποια στιγμή ε, ότι οι ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ασχοληθούν και με την κοινωνική πτυχή. Τι εννοείται, πώς το εννοείται. Δεχόστε τις ιδέες του συναδέλφου Σβόποτα και της Σοσιαλιστικής Ομάδας ότι λέμε ναι, όλοι οι νέοι πρέπει να έχουν μια προοπτική και θα το φροντίσουμε αυτό. Θέλετε ε, μισθού σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη που δυναμικά θα προσαρμόζονται στην οικονομική ανάπτυξη. Το θέλετε αυτό. Λέτε χρειάζεται ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής οι υπηρεσίε σας είπαν ότι δεν έχει αυτό καμία σχέση με επενδύσεις και θα γίνει μόνο με διαστατικές αλλαγές. Γι' αυτό το μνημόνιο συνεννόησης είναι τόσο μετριοπαθές. Πού είναι ο διάδρομος επενδύσεων που είχε απόφαση. Αν δεν πείτε ναι στις να, επενδύσεις λέτε ε, όχι και στην ανάπτυξη. Τελείωσε πια ο χρόνος των λόγων. Πράξεις χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπούλμαν και για τους υποστηριχτές που έχετε εδώ κοντά σας. Ο κύριος Σεφλίν για δύο λεπτά. President, um... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εγκρίνει την υποψηφιότητα της Σερβίας έχει διτή σημασία. Για την ίδια της Σερβίας την ουσία σημειώνει το τέλος θα έλεγα της μεταπολεμικής περίοδου και ταυτόχρονα οι Σέρβοι ε, θα πάψουν να αντιμετωπίζονται αρνητικά σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Η Σερβία μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα ότι έχει επιστρέψει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό έχει και μακροπρόθεσμη σημασία. Θα έλεγα αν θέλουμε να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή θα πρέπει να γίνει μαζί με τη Σερβία. Η Σερβία πρέπει βέβαια να κάνει ακόμα περισσότερα βήματα στα πλαίσια της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Αν δεν γίνει αυτό τα Βαλκάνια θα είναι εύκολο τόπος για τις διεθνείς μαφίες. Είναι σαφές επίσης ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει πιο αργά από ό,τι στο παρελθόν, αλλά δεν έχει σταματήσει. Αυτό έχει σημασία για τα Βαλκάνια. Και παρά την οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει τη σταθερότητα στις γειτονικές της περιοχές. Ο δικός χάρτης ε, τον οποίο ακολουθούμε νομίζω έχει σαν στόχο να πετύχουμε. Ε, οι στόχοι αυτοί βέβαια θα εξαρτηθούν από την προσπάθεια ε, που γίνεται να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση. Οι αποφάσεις οι τελευταίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να συμβαδίζει με την αναγνώριση της σημασίας της οικονομικής ανάπτυξης τη απουσία οικονομικής ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πολύ λιγότερο ελκυστική και δεν θα μπορεί να επηρεάζει έστω και με τον τρόπο που το κάνει. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Καλφίν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο πρόεδρος Μπαρόσο είπε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς σταθερότητα. Όμως αυτό είναι κοινοτυπία. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και σταθερότητα χωρίς μια οικονομία η οποία να αναπτύσσεται και να είναι δυναμική. Το πρόβλημα το οποίο να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι ότι τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση είναι διαφορετικής κατηγορίας, είναι διφορούμενα μέτρα έχουμε καταρχάς φορολογικά μέτρα και, ε, τα οποία έχουν όμως σοβαρές κυρώσεις και ε, προβλήματα, συνέπειες. Από την άλλη πλευρά για την ανάπτυξη ακούμε ωραία λόγια χωρίς όμως ουσία. Το αποτέλεσμα είναι σαφές και είχα την ευκαιρία να το δω και με τους σοσιαλιστές ε, συναδέλφους μας στην Ελλάδα. Διότι δεν υπάρχει η ικανότητα από πλευράς της, πολιτι... της ε, οικονομικής πολιτικής να ε, γίνει σεβαστό το χρέος. Και τι χρειάζεται, ποια είναι η λύση, είναι διαφορετικέ αλλαγές, ε, μια πιο ισχυρή, ένας πιο ισχυρός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος να στηρίζεται στους ιδίους πόρους και ένας δίκαιος καταμερισμός του χρέους. Για δύο λεπτά ο Στόλογιαν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είμαι και ικανοποιημένος και χαρούμενος για τον τρόπο με τον οποίο συνεισέφερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της κατάστασης των κρατών μελών που έχουν ε, υπερβολικό βάρος από το χρέος. Αυτό διεκπαιρεώθηκε. Αλλά είμαι απογοητευμένος γιατί η Ρουμανία και η Βουλγαρία παραμένουν εκτός Σέγγεν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρόλο που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ένταξη τους στη συμφωνία αυτή. Και τώρα πραγματικά είναι πρόβλημα μία χώρα αντιτίθεται στην ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Και δεν είναι τυχαίο κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω στην Ολλανδία ένα μικρό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση ανέλαβε και την πρωτοβουλία να ε, ξεκινήσει έναν ιστότοπο που αποτελεί προσβολή όσο και ύβρι στις ευρωπαϊκές αξίες και ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ένωσης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ε, Συμβουλίου ήταν χλιαρή δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες, πιστεύω, σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι κατά των ευρωπαϊκών αξιών και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απόγευμα να προχωρήσει σε μέτρα για να καταδικάσει αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ποδηματά για ένα λεπτό παρακαλώ. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ενθαρρυντικό το γεγονό ότι όλοι αναγνωρίζουμε πλέον ότι η μονομερής αιμονή στα μέτρα δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί να βγάλει ούτε την Ελλάδα από την κρίση ούτε την Ευρώπη από τη στασιμότητα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε αποφάσεις δεσμευτικές και έργα, δεν αρκούν τα λόγια και οι ευχές και για να είμαστε συγκεκριμένοι και πιστικοί απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες μπορούμε και πρέπει να συνδέσουμε συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα όπως ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή το ευρωομόλογο με το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο. επιτρέψτε μου ωστόσο να απευθυνθώ και στις διάφορες πυθίε που υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα και εκτός και που μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας και της ευημερίας του ελληνικού λαού για έξοδο της ελλάδας από το ευρώ και βεβαίω ο καθένα μπορεί να έχει την άποψή του σε αυτό το κοινοβούλιο έχουμε κατακτήσει την δημοκρατία προ θεού όμω μην επικαλείστε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. ο ελληνικό λαό με μια τεράστια πλειοψηφία του 70% έχει ταχθεί υπέρ τη παραμονή τη χώρα του ευρώ και δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιεί κανεί τι δικέ του δυσκολίε για να εξυπηρετούνται συμφέροντα διάλυση τη ευρωζώνη που προωθούνται συστηματικά από ορισμένου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να θυμίσω ε, και να παρακαλέσω τους ομιλητές να τηρούν το χρόνο τους. Αλλιώς αν μιλάτε όλοι 10 δευτερόλεπτα παραπάνω δεν θα ψηφίσουμε πριν τις 2. Ο κύριος Ρανζέλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας Ε, στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ε, γιατί, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε το Συμβούλιο. Δεν είναι ιδανικά τα, τα μέτρα τα οποία θα τις υιοθέτησαν, αλλά είναι εφικτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πλέον ε, η επικρατεί ένα μεγάλο ρεαλισμό από ότι πριν από τρει ή έξι μήνες. Και πάρα πολλέ χώρε έχουν προχωρήσει σε προσπάθειες ε, σταθεροποίηση, έχουν βάλει μια τάξη ε, στα δημόσια οικονομικά τους και Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να επανακτήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς ε, ε, οικονομικές αγορές για να μπορέσουμε να καλύψουμε τον ε, χαμένο χρόνο. Και πιστεύω ότι έχουν δοθεί κάποιες εγγύησεις από πολλά κράτη και πιο συγκεκριμένα από την Πορτογαλία για την οποία μιλάω για την ε, για το δημόσιο χρέος και είμαι σίγουρος ότι και με τη νέα συμφωνία που υπογράφηκε από τους 25 ε, θα μπορέσουμε στο επόμενο Συμβούλιο τα νέα να είναι πολύ πιο θετικά. Γιατί πιστεύω ότι με βάση όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλουμε θα υπάρξει ανάπτυξη. Και ε, επίσης πιστεύω ότι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους οχούς και τους πλούσιους θα δώσει τα καρπούς. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Ρότσεκ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η τσεχική δημοκρατία υπό την ηγεσία της γύρω, σκεπτικιστικής κυβέρνησης και τον ευρώφοβο πρόεδρο που έχει δεν υπέγραψε το δημοσιονομικό σύμφωνο. Ως πολίτης της τσεχικής δημοκρατίας πρέπει να πω ότι είναι σφάλμα. Και γεωγραφικά και πολιτικά η τσεχική δημοκρατία αλλά και οικονομικά είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι ζωτικό τη συμφέρον από πλευρά ασφάλειας, πολιτικής και οικονομικής να συνεισφέρει πλήρω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συμπεριλαμβανομένης βεβαίω, οποιασδήποτε ε, ολοκλήρωσης ε, νομισματικής και δημοσιονομικής. Αυτή είναι η άποψη των Τσέχων σοσιαλδημοκρατών και αυτή είναι και η άποψη της πλειονότητα της τσεχική κοινωνία, που όπω γνωρίζετε σε δημοψήφισμα ρητός εξέφρασε ε, την ε, άποψή της ότι ήθελε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως το Δημοσιονομικό Σύμφωνο δεν είναι πανάκια. Όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι προηγουμένω, θέλουμε να έχουμε περισσότερη απασχόληση, περισσότερε επενδύσει, περισσότερη κοινωνική πολιτική. Αλλά η δημοσιονομική ευθύνη είναι εκ των όνου κάνευ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα παρακαλώ η κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, οι αποφάσει του Συμβουλίου δείχνουν ότι υπάρχει πρόοδο και δρόμο που έχει διανυθεί Βεβαίω υπάρχει συχνά κακοφωνία και ευχή όλων μα είναι να υπάρξει μείωση των εντάσεων Όμω μαγικέ λύσει και ευχάριστε δεν υπάρχουν. πρέπει να υπάρξουν αποφάσει σε επίπεδο Ευρώπη και εντό των κρατών μελών. οι διαρθρωτικέ αλλαγέ θα βοηθήσουν ιδιαίτερα σε χώρε όπω η δική μου. μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί η κρίση του σήμερα και θα υπάρξει ελπίδα για ανάπτυξη. το δημοσιονομικό σύμφωνο το ευρωπαϊκό εξάμεινο και αποφάσει για την ενίσχυση τη απασχόληση μπορούν και πρέπει να γίνουν οδηγοί για την περαιτέρω πορεία. η ευρώπη διαθέτει και την ιστορία και την επίγνωση του συμφέροντος των ευρωπαίων πολιτών ώστε να μην επιτρέψει επί πολύ να την καταβάλει η οικονομική κρίση. το ιδεολογικό περιεχόμενο της κοινή μας προσπάθειας μαζί με τις προσπάθειες για ανάπτυξη θα δώσουν ελπίδα στους νέους της ευρώπης. το θέμα είναι οι θυσίες να έχουν πραγματικό αντίκρισμα. θέλω να σας τονίσω ότι ο ελληνικός λαός υποβάλλεται σε πολύ μεγάλες θυσίες γιατί δεν είναι διατεθειμένος να διακυβεύσει την παρουσία του στην ευρωπαϊκή ένωση και στο ευρώ ό,τι και αν ισχυρίζονται οι διάφορες κασάνδρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και ε, για το χρόνο που τηρήσατε. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Γκόμες παρακαλώ. O pacto orçamental assinado há dias é a demonstração que Το δημοσιονομικό σύμφωνο που γράφηκε πριν από μερικέ μέρε δείχνει ότι η ανάπτυξη και η ανεργία ακόμη είναι στο περιθώριο του ενδιαφέροντο των Ευρωπαίων ηγετών. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, αποτελούν την πηγή τη απασχόληση, και κυρίως των νέων, όπω είπε ο κ. Μπαρόζο. Εάν αυτό ισχύει λοιπόν, βλέπω ότι είναι σκανδαλώδηση η αδιαφορία των κρατών και κυρίως της ε, άρνησης πιστώσεων για την ανάπτυξη και, της, ε, και την απασχόληση στις χώρες που δανειοδοτούνται. Γιατί τα χρήματα αυτά πάνε στις τράπεζες αλλά δεν προσφέρουν οι ίδιες οι τράπεζες στη συνέχεια στον ενδιαφερόμενο πιστώσεις με, με ενδιαφέροντα κονδύλια. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αναφέρεται μόνο σε δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας, δεν δίνει όμως λύσεις για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι νέοι Ευρωπαίοι τώρα μεταναστεύουν, πάνε στο εξωτερικό. Στην ε, Πορτογαλία με ποσοστό ανεργίας των νέων πάνω από 35% η κυβέρνηση παραμένει απόλυτα αδρανής και δεν είναι σε θέση να προσφέρει ε, ελπίδα και προσδοκίες στους νέους. Δεν τρέπονται, δεν εσχύνονται. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βόρτμαν Κόλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε φτάσει σε καμπή. Φαίνεται ότι οι αγορές επανακάμπτουν όπως και η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, έχει δίκιο ο κύριος ε, Ρόμπαϊ, ο πρόεδρος. Και τώρα θα πρέπει να ξανάρθουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας και να δημιουργήσουμε ένα επενδυτικό κλίμα με εμπιστοσύνη. Οι επιχειρήσει έχουν πολλά χρήματα στι τράπεζε και οι ιδιώτε επενδυτέ δεν τολμούν να επενδύσουν. Αν ε, επανακάμψει η εμπιστοσύνη, θα έρθουν και οι επενδύσει για να κινητοποιηθεί και η ανάπτυξη τη οικονομία. Τα πάντα όμω θα εξαρτηθούν εάν ε, από το ΕΑΝ όμω θα δώσουμε συνέχεια στα λόγια μας με έργα. Ε, έγινε λόγος από τον Πρόεδρο για τη στρατηγική ανάπτυξη. Μα υπάρχει στρατηγική για το 2020, για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα πρέπει όμω να τα υλοποιούμε αυτά. Και αυτό θα γίνει μόνο αν το κάνουμε εμείς, ε, δεν θα πρέπει ο καθένας να ε, επιρρύπτει τι ευθύνε των άλλων. Η Κομισιόν στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο στα κράτη-μέλη. Ε, είναι εξαιρετική η επιστολή των 12 ηγετών και ε, λέει τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ας πούμε σε θέματα ε, φορολογίας, σε θέματα υλοποίησης στρατηγικής το 2020, στον ίδιο τους τον προπολογισμό, με αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, με προσπάθειες στην παιδεία και στις άλλες υπηρεσίες. Έτσι θα βγούμε από την κρίση και μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε τα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής σήμερα το πρωί και του Προέδρου του Συμβουλίου είναι πολύ πιο ανησυχητικά από το κείμενο της, ε, του Συμβουλίου, τα συμπεράσματα ε, του Συμβουλίου, διότι πολλά λόγια χωρίς κάτι συγκεκριμένο που είναι η οικονομική σταθερότητα και τα απαραίτητα μέτρα για να τα υλοποιήσουμε. Δεν θα τονίσω εγώ την σημασία αυτής της κατευθυντήριας γραμμής, αλλά προφανώς η ανάπτυξη, η κατάσταση πολλών εκατομμυρίων πολιτών θα επιδεινωθεί στην Ευρώπη και υπάρχει μια επαναχώρηση της οικονομίας ε, των χωρών μας ε, που είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό τους επόμενους μήνες αν δεν υπάρχουν επενδύσεις ε, και αν δεν αντιστραφεί αυτή η τάση θα έχουμε τεράστια κοινωνικά προβλήματα επομένως τα ευρωομόλογα και οι φόροι για τις συναλλαγματικές, για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανταλλαγές, συναλλαγές για τις συναλλαγές δεν πρόκειται να φτιάξουν την κατάσταση. Άλλα χρειάζονται για να, βελτιωθούν, ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για ένα μισό λεπτό, κύριος Χόικμαρκ. Κύριε Πρόεδρε, Yeah. η ευρωπαϊκή οικονομία, οικονομία υπέφερε από πολύ λίγες δημόσιες δαπάνες και πολλέ επενδύσει δεν θα είχαμε προβλήματα. Το λέω αυτό γιατί η συζήτηση που ακούστηκε εδώ δίνει την εντύπωση ότι με αύξηση των δημοσίων δαπανών, με αύξηση των ελλημάτων θα μπορούσαμε να επιτύχουμε οικονομική, ε, κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη. Ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Οι ανεξέλεγκτε δημόσιε δαπάνε, τα μεγάλα δημόσια ελλείμματα υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και οδηγούν σε αύξηση των επιτοκίων. Όσοι λοιπόν πιστεύουν ότι η αύξηση των δημοσίων δαπανών αποτελεί τη λύση στα προβλήματά μας, καλό θα κάνει να κοιτάξει γύρω του και να δει τα προβλήματα κατάματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο για ε, όθηση στην οικονομία και είναι πολύ σημαντικό εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιληφθεί ότι ο δρόμος, η οδός για την κοινωνική συνοχή ή και την κοινωνική ασφάλεια δεν βαίνει παράλληλα με την ε, οικονομική ανάπτυξη, με τον δρόμο για την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη, οι νέες θέσεις εργασίας είναι η λύση που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας κατά τρόπο ικανοποιητικό για τους πάντες. Και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις για την ιστορική αγορά, στις μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα στα κράτη-μέλη και να επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο αυτό να καταστεί μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πλουμ. Πρόεδρε, έλαβα μέρος στη συζήτηση για τα συμπέρασματα του Συμβουλίου και διαπιστώνω, ναι, συμφωνώ ότι χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα και ανάπτυξη και για να το επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ξεκάθαρα δημοσιονομικά σχέδια και να αναζητήσουμε τους πόρους εκείνους που προσφέρουν το δυναμικό για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Διότι πολλοί είναι οι πολίτες και κυρίως οι νέοι και οι γυναίκες που χρειάζονται μια θέση εργασίας και πρέπει αυτές τις θέσεις να τις δημιουργήσουμε. Άρα λοιπόν... Εάν αυτή η οδηγία για την εξοικονόμηση πόρων που ανέφερε ο κύριος Μπαρόσο που έχει ε, παραμείνει σε αδιέξοδο επίπεδο Συμβουλίου γιατί δεν προχωρεί. Γιατί δεν προχωρεί επίσης ε, η πρόταση για την άδεια ε, τοκετού. Ελπίζω λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό και ελπίζω βεβαίω ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα γίνουν μέλη του Σέγγεν. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για μισή λεπτό κύριο Κέλαμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης θα μπορούσε να είναι τώρα ήρθε η ώρα της, εφαρμογής. Ήρθε η ώρα που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα βασικά προβλήματα βέβαια είναι ε, οι απαιτήσει οι επιταγές του Συμβουλίου. Δηλαδή, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα απαραίτητα, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια ανάπτυξη, θα πρέπει να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ευνοήσουμε την απασχόληση των νέων. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, η ενιαία αγορά παραδείγματο χάρη. Ο κύριος Μπαρόζο χρησιμοποίησε μια άλλη ε, έκφραση, η οποία είναι πολιτικά ορθή. Εμβάθυνση της ε, ενιαίας αγοράς. Ε, σήμερα είναι η ζήτησε και ο κύριος Δόλο να επωφεληθούμε για την επέτειο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς με την προσπάθεια να την ολοκληρώσουμε, να την εμβαθύνουμε. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να ε, ξεφορτωθούμε αυτόν τον προστατευτισμό ο οποίος ε, τα τα τελευταία χρόνια έχει υποσκάψει την προσπάθεια της Ευρώπης για ανάπτυξη και έχει υποσκάψει επίσης και την οικονομική της ε, αξιοπιστία. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Η ικανοποίηση για, την, για το ότι ξεφύγαμε από τον κίνδυνο βέβαια είναι πραγματικός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα λάθη τα οποία κάναμε τα τελευταία χρόνια. Και θα δεν θα πρέπει η ευχαρίστηση αυτή να μας εμποδίσει να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία δεν επέλυσε η, τελευταία, η στρατηγική των τελευταίων μηνών τα μέτρα λιτότητας, ο περιορισμός των μισθών δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν είναι ούτε από οικονομικής, ούτε από κοινωνικής, ούτε από οικονομικής πλευράς βιώσιμα μέτρα ε, οι ελληματικές δαπάνες δεν βοηθούν. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια, ε, ε, μια μεγαλύτερη προσπάθεια για επενδύσεις και είναι εφικτό κάτι τέτοιο αντιμετωπίζοντας και τις μακροοικονομικές προκλήσεις και μέσω τεράστιων επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργώντα ένα σύστημα ενιαίας διαχείρισης των των ελλημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει η να, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο από το 2014 και να υπάρξει μια πραγματική οικονομική κυβέρνηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γουαλτιέρη. Για ένα λεπτό και 30 το λόγο κύριος Κάραστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. ο, η σύνοδος κορυφής ούτε δραματική ήταν, ούτε έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και περιγράφεται ως ε, καλύτερο συμβούλιο από τα προηγούμενα. Ίσως αν δεν είχαμε τόση σκηνοθεσία και τόση ε, φασαρία να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Εκανοποίηση ε, για τα οικονομικά και καλό ήταν που δεν είχα συνεννοηθεί προηγουμένως η κυρία Μέρκε με τον κύριο Σαρκοζή και επικεντρωθήκαμε στη ε, συνεδρίαση την ίδια αντί να κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει κυρίε και κύριοι να επικρίνουμε λιγότερο ένα τον άλλον και να δρούμε περισσότερο. Ωραία επιτέλους έχουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο, έχουμε ε, νομοθεσία για τις μικρές επιχειρήσεις, για την ενιαία αγορά, έχουμε τη στρατηγική για το 2020, ας τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Έχουμε και το ε, τεστ για τις μικρόμεσαίες, θα πρέπει να το κάνουμε τη δοκιμή αυτή και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ε, τα μέτρα και τα μέσα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να τα αξιοποιήσουν για τους ιδίους πόρους για να έχουμε και αποτελεσματικότητα πολιτική αλλά και αξιοπιστία. Γνωρίζουμε ότι αυξάνεται ο μηχανισμό σταθερότητας. Ας μην αναβάλουμε τις αποφάσεις, ας τις εκτελέσουμε. Το κοσυφοπαίδιο δεν είναι πρόβλημα της Σερβίας θα πρέπει ε, τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει το γοσυφοπέδιο να το πράξουν. Ε, λοιπόν, ας ε, δρούμε περισσότερο και ας επικρίνουμε ένα τον άλλο λιγότερο. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the και πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν θα κερδίσω κανένα βραβείο του πιο δημοφιλούς πρόεδρου. Έχουμε πέντε λεπτά. Είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, άρα θα δώσω το λόγο σε πέντε ομιλητές από ένα λεπτό στον καθένα. Δεκαπέντε όμως έχουν ζητήσει. Παρακαλώ την κατανόησή σας, ένα στους τρεις μόνο. Για να προετοιμάζεστε και ψυχολογικά με τη σειρά. Μαρσέγεφ, Κούκοβιτς, Ταμπάιτζη, Λούχαν, Λόπες Αγγιλάρ και τελευταίος ο κύριος Μπρόνς. Για ένα λεπτό η κυρία Μαρσέγεφ πρώτα. Η οποία Απουσιάζει. Α, όχι, δεν. Ε, ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μιλούν για λιτότητα, για εξοικονόμηση πόρων και ανάπτυξη. Όμως με τόσα εκατομμύρια νέων ανέργων είναι απολύτως απαραίτητο να ε, ενθαρρύνουμε, να εκπαιδεύσουμε και να εξοπλίσουμε τους νέους μας έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται και με την επιχειρηματικότητα. Γιατί το να έχει κανείς ιδέες μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή αρχή χωρίς όμως την υλοποίησή της, χωρίς θάρρος για να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και άρα, σε αυτή την εποχή της μεγάλης ανεργίας, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό πνεύμα, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση των νέων μας, έτσι ώστε να τολμούν να ε, γίνονται επιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενοι και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους μόνο. τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταμπάζου, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Είναι η πρώτη ευκαιρία μετά από χρόνια ε, που ε, το Συμβούλιο δεν έδρασε πυροσβεστικά, αλλά η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Είναι σε κίνδυνο η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή την κλιμάκωση του χρέους χωρίς οικονομική ανάπτυξη. Πολλά υπόθηκαν, έγινε λόγο για την ανάπτυξη της ενιαίας ιστορικής αγορά τα ευρωομολόγα όσο γίνεται συντομότερο και άλλα πολλά, αλλά εκτός από αυτό χρειάζεται και ένα γενικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που να βοηθάει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να αναπτύχθει πραγματικά η Ένωση. Από την άλλη υπάρχει και βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα με τη λειτουργία του ευρώ. Διαπιστώνουμε ότι ως κοινό νόμισμα ενιαίο το ευρώ δεν προσφέρεται για χώρες που έχουν οικονομίες με διαφορετική ανταγωνιστικότητα. Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν δυσκολίες οικονομικές αυτές οι χώρες και είναι κοντά στην κρατική ε, χρεοκοπία και πτώχευση. Αυτό δεν είναι μόνο ε, ε, λάθο και φταίξιμο των κυβερνήσεων, αλλά τη κοινή αποτυχία του ευρώ. Γι' αυτό θέλει μεταρρύθμιση οπωσδήποτε και του ευρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Λούαν, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Σέγγεν ως χώρος του Σέγγεν αντιμετωπίζει την ε, εχθρική στάση της Ολλανδίας η οποία παρεμποδίζει την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Οι κάτω χώρες λοιπόν έχουν λάβει μια απόφαση η οποία οδηγεί σε καθυστερήσεις ως προς την έγκριση της ε, πρόσβασης, της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Και έτσι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ισότιμες ευθύνες ίσες ευθύνες βλέπουμε ότι δεν, έχουν, δεν απολαμβάνουν των δύο δικαιωμάτων ε, και προνομιών όλα τα κράτη-μέλη. Ορισμένοι λοιπόν φιλόδοξοι ηγέτες ορισμένων πολιτικών κομμάτων, ορισμένων κρατών στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης υπονομεύουν ε, την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενότητας, την Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δυνατότητα της λαμβάνει αποφάσεις. Και γι' αυτό ζητώ κάθε αρμόδιο όργανο να εντοπίσει και να υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμβάλλει στην επέκταση του χώρου Σέγγεν. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριος Λόπες Αγγιγιάρ, ένα λεπτό. Επανειλημμένα μίλησα για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για να μιλήσω για άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης ούτε την καταπολέμηση των οικονομικών ε, ανισορροπιών αλλά έχουν να κάνουν με τα θεμέλια τα ίδια και το λόγο ύπαρξη Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κοινότητα δικαίου και το ξαναλέω για άλλη μια φορά σε σχέση με τα τωρινά συμπεράσματα για τα θέματα ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης και την ελεύθερη κυκλοφορία στο Σέγγεν. Γιατί το Κοινοβούλιο τον Ιούνιο ψήφισε τη διεύρυνση του Σέγγεν προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και σύμφωνα με τις συνθήκες ε, πρόσβασης το 2005 είχαν κάποια κριτήρια και κάποιες προϋποθέσεις. Και το Συμβούλιο θεώρησε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι δύο χώρε, Αλλά και πάλι ανέβαλε την απόφαση και την παρέπεψε το Σεπτέμβριο του 2012 στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Το Κοινοβούλιο ελπίζει να υλοποιηθεί αυτή η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που πληρούν τα κριτήρια για να μπουν στη ζώνη Σέγγεν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει. Δεν συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση αυτά που ακούμε στη γαλλική προεκλογική εκστρατεία που απειλούν να επαναφέρουν τα εσωτερικά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος ε, δεν μας έχει εμπιστοσύνη και ακολουθεί τον αντίστοιχο, τον δρόμο από αυτό που επιθυμούμε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Μπρόνς. Ε, Η συνθήκη για τη δημοσιονομική πειθαρχία δεν σχετίζει την εφημερία των υπογραφώντων με την εφημερία του ευρώ και της ζώνης του. Απλώς επιβάλλει έναν ε, στενό κορσέ δημοσιονομικό στα κράτη της ευρωζώνης. Αναφέρεται βέβαια στο κρατικό χρέος, αλλά μόνο με δικτατορικές ε, επιταγές και όχι με δημοκρατικές λύσεις. Φέρνει δε σε μια ε, απεργία πείνα ουσιαστικά τα κράτη της ε, Νότιας Ευρώπης με πολύ μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, με ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στον προπολογισμό, με αναργία και επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων τα κράτη του ευρώ, τα κράτη αυτά μάλλον της Ευρώπη, θα πρέπει να αποχωρήσουν από το ευρώ και η αποχώρηση αυτή αποτελεί τη μόνη λύση για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Για να μπορούν να δανείζονται σε πολύ πιο φθηνού όρου, πιο οικονομικού όρου, πρέπει να φύγουν από το ευρώ. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα ο κύριο Σεύκοβιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι πολλά από τις ερωτήσεις έχουν πάρει μια απάντηση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα τα οποία έθιξαν οι περισσότεροι από τους ομιλητές. Οι εργασίες, η ανάπτυξη, και το πού θα βρούμε επενδύσεις για να χρηματοδοτήσουμε τις δράσεις μας. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι η ανεργία και κυρίως η ανεργία των νέων είναι μία από τις πέντε ε, προτεραιότητές μας που θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας φέτος. Είναι το αποτέλεσμα ενός, ε, μιας έρευνας που κάναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε και σε κάθε ε, πρόγραμμα των, κρατών μελών το θέμα αυτό να έχει την ύψιστη προτεραιότητα διότι είναι ε, προφανές ότι είναι σημαντικό για όλους μας να έχουμε θέσεις απασχόλησης και θέλουμε να έχουμε και ανθρώπους που να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουμε μια, εργασία, μια αγορά εργασίας η οποία να λειτουργεί καλύτερα και να ε, δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της οικονομίας, αλλά θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας και στους τομείς όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, επικοινωνία, ε, τεχνολογία της πληροφορικής, IT γενικότερα Επίση ε, Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τα εμπόδια τα οποία ακόμα εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και την εργατική δυναμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους που αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες πιέσεις στην αγορά εργασία. Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε 7,5 εκατομμύρια νέους που δεν είτε εργάζονται είτε δεν καταρτίζονται είναι ένα από μία από τις προθέσεις ε, της ε, Κομισιό να έχουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις τις οποίες θα εφαρμόσουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης θέλουμε να υπάρχει μία εγγύηση για τους νέους Δηλαδή ότι οι νέοι από τη στιγμή που θα τελειώσουν τις σπουδέ τους θα έχουν την εγγύηση είτε θα βρούνε, να βρουν θέσεις απασχόλησης είτε να περάσουν επαγγελματική κατάρτιση ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των ε, νέων στην Ευρώπη. Επίσης θα βελτιώσουμε τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τα, τους ενδιαφερομένους να βρούνε μια δουλειά. Θα πρέπει να προτείνουμε ε, κάποια προγράμματα τα οποία θα ε, ε, επιτρέπουν στα κράτη-μέλη, θα επιτρέπουν στους νέους να βρίσκουν δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Τώρα, από το πού θα βρούμε τα χρήματα, από πού θα βρούμε τις επενδύσεις, τώρα που περνάμε μια περίοδο λιτότητας, περίοδο κρίσης. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τα όσα δραματικά ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Αν ε, μιλήσουμε για θέσεις νέες απασχόλησης ε, και για επενδύσεις, ε, πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε καταρχάς την χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Έχουμε 21 δισεκατομμύρια στο κοινωνικό ταμείο και άλλα 21 δισεκατομμύρια από, το, από τον Διαρθρωτικό Ταμείο δεν έχουν δαπανηθεί. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βρούνε κάποιες προτεραιότητες. Ε, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν θέσεις για τους νέους και για τους νέους αλλά και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ακούστηκαν διάφορες ιδέες <clears throat> για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και άλλο εισόδημα ή και άλλες επενδύσεις. <clears throat> Νομίζω ότι ε, συμφωνούμε απόλυτα από αυτού, διότι η Κομισιό και το ξέρετε ε, και με την ε, πρόταση για τον φόρο των οικονομικών συναλλαγών ότι εμείς ε, αυτό θέλαμε, το είχαμε προτείνει. Αλλά χρειάζεται όμως ομοφωνία για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Επίσης ε, για, προχωράμε και για τα project για τα ομόλογα ε, γιατί οι αρχικές μας ε, έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν προοπτικές. Έχει γίνει προσπάθεια μόχλευσης και θα βρούμε τα χρήματα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την ιδιωτική αγορά. Αυτά είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για υποδομές, για το ICT, να προσφέρουμε θέσεις απασχόλησης έτσι ώστε να βελτιωθεί και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ξέρετε ότι υποστηρίζουμε τους ιδίους πόρους και σε κάθε συνάντηση που λαμβάνει η χώρα με τα κράτη-μέλη το θέτουμε το θέμα και εσείς παίρνετε τις πληροφορίες βέβαια από τους δικούς σας διαπραγματευτές. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση. Αλλά πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε πιο διάφανο προϋπολογισμό θα πρέπει να ε, έχουμε ε, ιδίους πόρους, ισχυρούς ιδίους πόρους για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα έλεγα και κάτι άλλο ακόμα. Ε, αν εξετάσετε την πολιτική επενδύσεων, ένα καλύτερο, το καλύτερο επενδυτικό εργαλείο στην Ευρώπη είναι ο προπολογισμό. πού θα βρείτε αλλού έναν προπολογισμό του οποίου το 94% επιστρέφει στα κράτη-μέλη και ενισχύει τα έργα και που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάζουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για, το, για την ενιαία αγορά και για την δυνατότητα να προχωρήσουν από ένα fast track τα, τα, κάποιες προτάσεις μας. Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης ε, και ανάπτυξη. Τώρα για την Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τον Σέγγεν. Ξέρετε ότι είναι σαφή η θέση της Κομισιόν. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στο Σέγγεν και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε ήδη αυτά τα δύο κράτη να ήταν μέλη του Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και για αυτό το σημείο τη ημερήσιας διάταξη. Απλώ ε, σα ενημερώνω για το επόμενο θέμα τη ημερήσιας διάταξη ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει